Colleagues, would you take your seat, please? Σας παρακαλώ να καθίστε στις θέσεις σας, αγαπητοί συνάδελφοι. Liebe Kolleginnen, liebe Αγαπητοί συνάδελφοι, συναδέλφοι σας καλωσορίζω στην πρώτη συνεδρία της Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Μία σύντομη συνεδρία πριν το καλοκαιρινό διάλειμμα. Και ξεκινώντας να καλωσορίσω τον Υπουργό Απασχόλησης ε, της Ιταλίας, τον Τζουλιάνο Πολίτη. Καλωσορίσατε κύριε Υπουργέ. Μας δίνετε, το, μας δίνετε τη δυνατότητα να συζητήσουμε αναλυτικά για, την, ε, για το πρόγραμμα της Ιταλικής Προεδρίας. Um να επιβεβαιώσω όμως καταρχήν την ημερήσια διάταξη και να κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις στην πλευρά του Προεδρείου. Στη ημερήσια διάταξη έχουμε αρχικά μια ανακοίνωση από τη δική μου την πλευρά, μετά ανταλλαγή απόψε με τον Τζουλιάνο Πολίτη, την παρουσίαση του προγράμματος της Ιταλικής Προεδρίας και μετά ασχοληθούμε με τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο σημείο 5 την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για τη συνεργασία, για την αποφυγή και την ε, επάταξη της αντίληψης εργασίας. Η επόμενη συνεδρίαση στη συνέχεια και έχουμε και τα λοιπά θέματα. Να κάνω κάποιες ανακοινώσεις από την πλευρά μου. Να σε ενημερώσω για το κλασικό καθεστώς. Έχουμε όλες τις γλώσσες, εκτός από τα φιλανδικά, τα ε, μαλτέζικα, τα κροάτικα. Συζητήσαμε ε, σε ομάδα συντονιστών το πρωί και συζήτησαμε και για τις γλώσσες που χρειαζόμαστε επιγόντως και αυτές, είναι τα δανέζικα, τα δανικά. Θα φροντίσουμε όλα αυτά τα θέματα να αντιθετηθούν. Δεν έχουμε περιπτώσει ε, που δεν ε, χρειάστηκε από την τελευταία συνεδρίαση. Στην αρχή κάθε περίοδου ε, να βγάζουμε μια οικογενειακή φωτογραφία και γι' αυτό σημειώστε την 3η Σεπτεμβρίου, 5 η ώρα, 5 Σεπτεμβρίου, 3 η ώρα, θα βγάλουμε σε αυτή την αίθουσα την αναμνηστική φωτογραφία. Είναι web stream τη συνεδρίαση. Θα είναι διαθέσιμη και ηλεκτρονικά στο διαδίκτυο μέσω της εφαρμογής e-meeting. Θα προσπαθήσουμε επίσης να μειώσουμε τη χρήση χαρτιού. Βλέπετε ένα εγχειρίδιο μπροστά σας που αφορά το e-meeting. Μπορείτε να τις πληροφορίες, όλα τα έγγραφα από τις εργασίες της Επιτροπής θα είναι διαθέσιμα σε αυτή την εφαρμογή. Κατά πέμπτον, Υπάρχει ένα πακέτο καλωσορίσματος για τα μέλη της Επιτροπής και αυτό θα είναι διαθέσιμο σήμερα σε αυτήν την αίθουσα σε όλες τις ε, χώρες, ε, σε όλες τις επίσημες γλώσσες, με συγχωρείτε. Σε περίπτωση που κάποιος ευρωβουλευτής δεν είναι παρόν μπορεί να το παραλάβει ο βοηθός του. Εκεί υπάρχουν πληροφορίες για ε, την εισαγωγή της εργασίας της Επιτροπής. αν χρειάζεται πληροφορίες για τον τρόπο λήψης αποφάσεων, μπορείτε να πληροφορηθείτε και από τα θεματικά τμήματα και από άλλες πηγές. Εδώ σας ε, παρουσιάζουμε μια γενική σύνοψη για την 8η κοινοβουλευτική περίοδο. Αυτό το Welcome Pack θα είναι θέσιμο και στο site και στο e-committee από σήμερα το απόγευμα. Πάμε στο σημείο 6 της ημερησίας διάταξης. Η σύνθεση της Επιτροπής έχει αλλάξει και πάλι. Ο Μάρκο Βάλι δεν είναι πλέον μέλος της Επιτροπής. Αντικαθίσταται από την κυρία Τσιάννα Μπεγίν, η οποία από σήμερα ανήκει στην Επιτροπή μας. Το πρωί είχαμε δύο συνεδριάσεις. Την πρώτη συνεδρίαση που ήταν το συντονιστών. Ασχοληθήκαμε με το σημεία. Και να σας πω για αυτά. Συμφωνήσαμε για το χρονοδιάγραμμα, για τις ε, εκθέσεις της πρωτοβουλίας, τις ε, γνωμοδοτήσεις και τις μελέτες που θέλουμε να εκπονήσουμε. Δεν έχουμε άπλετο χρόνο στη διάθεσή μας. Θέλουμε κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα εργασιών μας και να το ανακοινώσουμε. Και επίσης ε, συμφωνήσαμε ότι τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο θα έχουμε το τελευταίο την τελευταία διαθέσιμη ακροασή και που θα έχει να κάνει με το TTIP, με το TTIP και την απασχόληση ένα θέμα που ενδιαφέρει πολύ την ε, δημοσιότητα και γι' αυτό αποφασίσαμε σε μορφή ακρόασης ε, να το συζητήσουμε το θέμα εδώ. Θα προσφέρουμε και ένα workshop για τα νέα μέλη της Επιτροπής Απασχόλησης αλλά και για τους βοηθούς. Αυτό θα το διευκρινίσει όμως ε, η γραμματεία. Θυμάμαι και εγώ τις πρώτες μέρες ε, το ξεκίνημα της καριέρας μου εδώ και ξέρω ότι πολύ γρήγορα θα μπορέσετε να συνηθίσετε. Το πρωί έγινε και η πρώτη ε, συνεδρίαση του EGF Working Group. Η πρώτη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Θα το συγκάλε, θα συγκληθούμε και στην επόμενη συνεδρίαση για να αποφασίσουμε για ε, τον τρόπο συνέχισης των εργασιών σε αυτή την ομάδα. Τέλος, ζητήμε με μεγαλύτερη διαφάνεια από την πλευρά του Ευρωπαίου α, διαμεσολαβητή, από την πλευρά της Επιτροπής μας, για την Επιτροπή μας. Ε, ζητούν τα πρακτικά από τις συνεδριάσεις των συντονιστών θα είναι διαθέσιμα επομένω τα πρακτικά στην επόμενη συνεδρίαση για να εξασφαλίσουμε το μέγιστο βαθμό διαφάνειας. Ελπίζω να μπορέσουμε να συνεργαστούμε επιτυχώς στη συνέχεια. Αυτά ήθελα να πω από την πλευρά μου. Δεν ξέρω, Αντρέας, αν έχω ξεχάσει κάτι. Όχι, τότε λοιπόν μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 3 της μέρησιας διάταξης. Ανταλλαγή απόψεων με τον Υπουργό Τζουλιάνο Πολέτη. Ο λόγος σε εσάς να μας μιλήσετε για το πρόγραμμα της Τελικής Προεδρίας. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε αξιότιμοι ευρωβουλευτέ. Είναι για μένα πραγματικά μεγάλη τιμή να βρίσκομαι εδώ ανάμεσά σας ως Προεδρεύων του Συμβουλίου Έπσκρο Απασχόλησης Κοινωνικής Πολιτικής Υγείας και Κατανάλωσης. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της Επιτροπή σα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μελλοντική σα θετική συμβολή. Ως Προεδρεύων θα εργαστώ με ενθουσιασμό και αποφασιστικότητα προκειμένου να επιτύχουμε το στόχο μιας βιώσιμης ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς και προκειμένου να ενισχύσουμε τις θεμελιώδεις αρχές στις οποίες από κοινού βασιζόμαστε κατά τη διάρκεια της καθημερινής μας εργασίας, προκειμένου να επανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών προς την Ευρώπη μας. Ο ρόλος μας λοιπόν είναι πολύ σημαντικός και η πρόθεσή μου να αξιοποιήσω κάθε δυνατή ανταλλαγή απόψεων και συνεργασία που θα μπορώ να έχω μαζί σας στους κοινούς μας στόχους. Η Ιταλική Προεδρία έχει ως στόχο να προωθήσει μια περαιτέρω εξέταση όσον αφορά τις πολιτικές προτεραιότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αναπτύξει καινοτόμες προτάσεις που θα είναι σε θέση να επιφέρουν σημαντικέ βελτιώσει στι διάφορε διαδικασίε που ακολουθούμε. Θα εργαστούμε λοιπόν έχοντα ω βασικό κεντρικό στόχο την πρόθεση τη ανάπτυξη και τη απασχόληση και πιο συγκεκριμένα και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής σας, η Ιταλική Προεδρία θα επικεντρωθεί στις εξής πέντε προτεραιότητες. Πρώτον, απασχόληση των νέων. Δεύτερον, κοινωνική διάσταση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Τρίτον, καταπολέμηση της ένδυας, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Τέταρτον, κοινωνική οικονομία. Και πέμπτη προτεραιότητα, η πράσινη ανάπτυξη. Οι προτεραιότητες αυτές θα προωθηθούν στα πλαίσια της διαδικασίας αναθεώρησης της στρατηγικής Ευρώπη 2020, στην οποία η Ιταλική Προεδρία θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή, εμπλέκοντας όλες τις ομάδες του Συμβουλίου. Θα αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό επίσης και στο Συμβούλιο ΕΠΣΚΡΟ της 16 ης Οκτωβρίου στο Λουξεμβούργο και θα μας πασχολεί το ζήτημα αυτό και στην Τριμερή Κοινωνική Σύνοδο η οποία θα λάβει χώρα το πρωί της 23ης Οκτωβρίου του 2014. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω τώρα τη γενική προσέγγιση που θα έχουμε ως Ιταλική Προεδρία και η οποία βασίζεται σε τρεις σημαντικές πτυχές, σε τρία σημαντικά ζητήματα. Στόχοι, μέσα και διακυβέρνηση. Καταρχάς θα ήθελα να αφαιρθώ στο ζήτημα της διακυβέρνησης προκειμένου να τονίσω την αγκαιότητα να αναφερθούμε και στο πλαίσιο αυτό, στο ευρωπαϊκό εξάμεινο και στο πώς θα μπορούσαμε να το καταστήσουμε λίγο πιο λειτουργικό για την επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής Ευρώπη 2020. Τον Οκτώβριο θα δεξαχθεί μια ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων μεταξύ ΜΟΝ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να καταλήξουμε σε κάποιες προτάσεις που θα είναι σε θέση να ενισχύσουν την ανάληψη ευθύνης, την κυριότητα, την αξιοποίηση των μέσων επιτήρησης, την πρόθεση της συνεργασίας με τους βασικούς ενδιαφερομένους, καθώς επίσης και την αναθεώρηση ενός νέου χρονοδιαγράμματος, προκειμένου να καταφέρουμε να προωθήσουμε καλύτερα τις βασικές μας προτεραιότητες. Προσβλέπουμε λοιπόν στην συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και όσον αφορά την στρατηγική Ευρώπη 2020. Προσβλέπουμε λοιπόν στη δική σα επικοδομητική συνεργασία. Να περάσω τώρα σε κάποιε συγκεκριμένε προτεραιότητες, αυτές που ανεφέρθηκαν στην αρχή τη παρέμβασή μου. Πρώτον, απασχόληση των νέων. Αυτή είναι μία από τις πιο βασικές προκλήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα αποτελέσει αντικείμενο του, της, τρίτους, της τρίτης με συγχωρείτε, συνόδου κορυφής μετά το Βερολίνο και το Παρίσι που θα λάβει χώρα στο τέλος του Ιταλικού εξαμήνου. Θα επικεντρωθούμε κυρίως σε εκείνες τις μακροοικονομικές πολιτικές που μπορούν να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης καθώς επίσης και στο ότι θα πρέπει να καταλήξουμε σε μία ποιοτική και βιώσιμη εγγύηση για τους νέους καθώς αυτή μπορεί να αποτελέσει ένα μέσο αντιμετώπισης της ανεργίας στην Ευρώπη. Θα συζητήσουμε το ζήτημα αυτό επίσης και στο Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ του Δεκεμβρίου, που για πρώτη φορά θα διεξαχθεί παράλληλα με το Συμβούλιο Εκπαίδευσης και Νεολαίας. Δεν θα πρέπει όμως το ζήτημα αυτό της απασχόλησης των νέων να μας αποσπάσει από άλλες προτεραιότητες όπως η καταπολέμηση της μακροχρόνιας ανεργίας καθώς επίσης και το ζήτημα της απασχόλησης των γυναικών. Η δεύτερη σημαντική προτεραιότητα της Ιταλικής Προεδρίας είναι η ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Στην, στο άτυπο συμβούλιο που έλαβε χώρα την προηγούμενη εβδομάδα στο Μιλάνο, καταφέραμε να εμβαθύνουμε τη συζήτηση για το ζήτημα αυτό, την πολιτική μάλιστα συζήτηση, όσον αφορά το ζήτημα των αυτόματων σταθεροποιητών, εξετάζοντας τις προϋποθέσεις για τη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού συστήματος επιδόματος ανεργίας. Η συζήτηση η οποία έγινε για πρώτη φορά μεταξύ υπουργών και κοινωνικών εταίρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο δημιούργησε, αν θέλετε, μια πρώτη πραγματική ευκαιρία ανταλλαγή απόψεων για τι διάφορε επιλογέ που μπορούμε να έχουμε για αυτό το ευρωπαϊκό επίδομα ανεργία και μα επέτρεψε επίση να αξιολογήσουμε τι επιπτώσει ενό τέτοιου μηχανισμού σταθεροποίηση όσον αφορά τι πολιτικέ απασχόληση και όσον αφορά την σύγκληση των πολιτικών των κρατών μελών. Γνωρίζω το ζήτημα αυτό είναι ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο, αλλά ακόμα και στο πλαίσιο αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που ήδη έχει διεξάγει μια σχετική συζήτηση του τελευταίους μήνες πιστεύω ότι θα μπορέσει πραγματικά να συμβάλλει πολύ σημαντικά. Η άτυπη σύνοδος του Μιλάνου με φέρνει τώρα σε τρία σημαντικά επόμενα θέματα. Η καταπολέμηση της φτώχειας και ο κοινωνικό αποκλεισμό. Ιδίω σε συνάρτηση με την αθεώρηση στρατηγικής Ευρώπη 2020 πριν από τέσσερα χρόνια, μάλλον μετά από τέσσερα χρόνια από την έναρξη της στρατηγικής Ευρώπη 2020, βλέπουμε όλοι μας ποιε είναι οι δεινέ επιπτώσει και ποια είναι η διάρκεια τη οικονομική αυτή κρίση, η οποία μα έχει απομακρύνει από τον αρχικό μα στόχο να μειώσουμε κατά 20 εκατομμύρια τον αριθμό των απόρων και των κοινωνικά αποκλεισμένων μέχρι το 2020 προκειμένου να δώσουμε νέο έναυσμα και να αυξήσουμε τη φιλοδοξία της στρατηγικής αυτής, ιδίω για την καταπολέμηση της φτώχειας και τον κοινωνικό αποκλεισμό, στόχους που θέσαμε το 2010, νομίζω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε εκ νέου τους κοινωνικούς εκείνους δείκτες που χρησιμοποιούμε για να επιτύχουμε τους στόχους μας. Ξέρετε ότι οι δείκτες αυτοί ήταν αποτέλεσμα ενός πολιτικού την εποχή εκείνη συμβασμού. Στο Μιλάνο λοιπόν συζητήσαμε για τις προσπάθειε που θα πρέπει μονομένα αλλά και συλλογικά να καταβάλουν τα κράτη-μέλη για την καταπολέμηση τη φτώχεια, καθώ επίση και τα απαραίτητα μέσα τα οποία θα, θα μα επιτρέψουν να εντάξουν περισσότερο τι κοινωνικέ πτυχέ στι εθνικέ δημοσιονομικέ πολιτικέ. Το ζήτημα τώρα της κοινωνική οικονομίας είναι ένα ακόμα ζήτημα το οποίο μας απασχολεί και βρίσκεται ακόμα στο περιθώριο των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, ένα ζήτημα πάρα πολύ σημαντικό για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και για την υποστήριξη των συστημάτων πρόνοιας. Μέχρι στιγμής συναφερόμασταν κυρίως στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, θεωρώντας ότι ο τριτογενής τομέας είναι κατά κάποιο τρόπο περιττός ή περιθωριακός. Στο κέντρο όμως του πυλώνα αυτού βρίσκεται η πραγματική κοινωνία, οι πραγματικοί πολίτες, οι οποίοι σε καθημερινή βάση προσπαθούν να λάβουν δράση ο καθένας στη χώρα του για να καλύψουν ανάγκες τις οποίες δεν μπορεί ή δεν δύναται να καλύψει το κράτος. Με τους συναδέλφους μου λοιπόν θέλω να ξεκινήσω μια νέα συζήτηση για τα προβλήματα και τις προκλήσεις της κοινωνικής οικονομίας και ιδίως για το πώς θα μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε περισσότερο την οικονομία αυτή, η οποία με σίγουρος θα οδηγήσει στη δημιουργία περαιτέρων θέσεων απασχόλησης, ποιοτικών θέσεων απασχόλησης. Νομίζω ότι πρέπει να βαθύνουμε όμως και σε έναν άλλον τομέα. Ένα ζήτημα το οποίο μας απασχόλησε ήδη σε μια συζήτηση που είχαμε σε υπουργικό επίπεδο με τους Υπουργούς Απασχόλησης και Περιβάλλοντος στο Μιλάνο. Το ζήτημα δηλαδή της πράσινης ανάπτυξης δεν το έχουμε εκμεταλλευτεί ακόμα πλήρως το ζήτημα αυτό Σίγουρα υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι όσον αφορά την μετάβαση προς μια πιο πράσινη οικονομία, κίνδυνοι τους οποίους θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε για να αποφύγουμε οποιοδήποτε φαινόμενο ανεργίας το οποίο θα μπορούσε να προκύψει από την πράσινη αυτή ανάπτυξη. Θεωρώ ότι η συνεργασία των δύο θεσμικών μας οργάνων και στον τομέα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική προκειμένου να καταφέρουμε στη δύσκολη αυτή περίοδο για την Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθήσουμε μια βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς να σε εκθέσω τώρα πώς έχουν τα πράγματα όσον αφορά τα διάφορα εκκρεμή νομοθετήματα. Πρώτον, θα ήθελα να αφαιρθώ στην πρόταση απόφασης για την αδήλωτη εργασία. Η αδήλωτη εργασία είναι ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει ακόμα περισσότερο τόσο στον τομέα της πρόληψης όσο και στον τομέα του, της καταπολέμησης. Η λαθρέα δήλωτη εργασία έχει σαφώς επιζήμιες επιπτώσεις, κυρίως στις συνθήκες εργασίας των ατόμων, αλλά είχε ε, επιζήμιες συνέπειες και στο θεμητό ανταγωνισμό, καθώς επίσης και στο dumping το κοινωνικό, επίσης ε, όσον αφορά και τους δημόσιους προπολογισμούς. Η πρόταση λοιπόν απόφαση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει τη δημιουργία μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα προκειμένου να αυξηθεί η συνεργασία μεταξύ κρατών μελών σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να καταπολεμήσουμε αποτελεσματικά το σχετικό αυτό φαινόμενο. Η πλατφόρμα λοιπόν αυτή θα διασφαλίσει συνεργασία όλων των οργάνων ελέγχου καθώ επίση και τη συμμετοχή άλλων ενδιαφερομένων όπω για παράδειγμα οι εκπρόσωποι εργοδοτών και εργαζομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να ανταλλάξουμε βέλτιστε πρακτικέ, θα βελτιώσουμε τα εθνικά και κοινοτικά μέσα και θα καταφέρουμε να καταλήξουμε τελικά σε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές, όπως για παράδειγμα με τη δημιουργία ευρωπαϊκών εκστρατιών ενημέρωσης. Κινούμεθα ήδη ιδιαίτερα επικοδομητικά στο ζήτημα αυτό στο Συμβούλιο και πιστεύω ότι ήδη τον Οκτώβριο θα είχαμε καταλήξει σε κάποιον γενικό προσανατολισμό. Είναι σαφώς δύσκολο να κινούμεθα σε ένα κοινό πλαίσιο όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν νόμοι, συστήματα μέσα τα οποία αποκλίνουν πάρα πολύ από κράτος μέλος σε κράτος μέλος και βλέπουμε ότι τελικά κινούμεθα με έναν τρόπο τελώς διαφορετικό στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης Και το ίδιο το φαινόμενο αυτό παρουσιάζει πολλές διαφορετικές παραλλαγές. Ωστόσο, νομίζω ότι θα πρέπει να συμμετέχουν στην όλη διαδικασία όλα τα κράτη-μέλη, με τη δυνατότητα για το καθένα να συμβάλλει υποστηρίζοντας τα υπόλοιπα κράτη-μέλη στους τομείς εκείνους που έχει προχωρήσει περισσότερο και μπορεί λοιπόν να συμμετέχει το κάθε κράτος μέλος στις πρωτοβουλίες εκείνες που το αφορούν περισσότερο ή που είναι πιο συμφέρουσες γι' αυτό. Ελπίζω και πάλι ότι η Επιτροπή σας θα διορίσει σύντομα έναν εισηγητή για να καταφέρουμε έστω και άτυπα να ξεκινήσουμε μια ανταλλαγή απόψεων για την πρόταση αυτή απόφαση, για την αδήλωτη εργασία που είναι πάρα πολύ σημαντική. Ένα άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο πρέπει να μα απασχολήσει ταχύτατα είναι αυτό που έχει να κάνει με τον κανονισμό για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υπηρεσιών Απασχόλησης, το δίκτυο EURES. Γνωρίζουμε ότι το μέσο αυτό μπορεί να διευκολύνει την κινητικότητα των εργαζομένων, ζήτημα το οποίο μας απασχολεί όλος ιδιαιτέρως και στο οποίο αφιερώσαμε μια ιδιαίτερη συζήτηση στην άτυπη σύνοδο του Μιλάνου. Η ολοκλήρωση του δικτύου αυτού ΕΡΕΣ μπορεί να βοηθήσει επίσης στην καταπολέμηση της νανικής ανεργίας οι νέοι, όπως ξέρετε, κινούνται πολύ περισσότερο από τους υπόλοιπους και επομένως είναι καθήκον μας να διαθέσουμε προς τους νέους ε, τις απαραίτητες συνδευτικές υπηρεσίες υποστήριξης προκειμένου να συμβάλλουμε στην ανάπτυξή τους, τόσο προσωπική όσο και επαγγελματική. Το Συμβούλιο άρχισε ήδη να εξετάζει την πρόταση αυτή κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας και εμεί θα βασιστούμε στα πορίσματα της προηγούμενη λοιπόν Προεδρία προκειμένου να προωθήσουμε περισσότερε διαπραγματεύσει ελπίζοντα ότι θα καταφέρουμε πολύ σύντομα να καταλήξουμε σε συμφωνία στα πλαίσια του Συμβουλίου. Βέβαια, προφανώς υπάρχουν ακόμα και άλλα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να εξετάσουμε και να εμβαθύνουμε περισσότερο. Αλλά αυτό το οποίο με καθησυχάζει είναι ότι επί της ουσίας υπάρχει μια κοινή συνένεση όσον αφορά τους στόχους που πρέπει να προωθήσουμε και αναφέρομαι κυρίως στους στόχους εκείνους που έχουν να κάνουν με την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. Ελπίζω ότι θα καταφέρουμε λοιπόν να ξεκινήσουμε ένα επικοδομητικό διάλογο με την Επιτροπή σας. Αυτή τη στιγμή θα έχουμε πλέον και έναν για το δίκτυο EURES. Εν τέλει θα ήθελα να αναφερθώ και στην πρόταση οδηγίας για τους ναυτικούς, η οποία έχει ως στόχο να δημιουργήσει ένα ομογενές επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων των ναυτικών σε όλους τους χώρους εργασίας τους. Γνωρίζουμε ότι σαφώς υπάρχουν κάποιες ανησυχίες που έχουν να κάνουν με τις ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί η οδηγία αυτή να έχει για τον ανταγωνισμό του τομέα αυτού, του κλάδου αυτού σε διεθνές επίπεδο. Είμαι όμως πεπισμένος ότι με την κατάλληλη ανταλλαγή απόψεων θα καταφέρουμε να μετριάσουμε αυτές τις ανησυχίες. Ελπίζω ότι η Επιτροπή σας θα ξεκινήσει σύντομα την εργασία της για την πρόταση αυτή οδηγίας και από τη δική μου την πλευρά, από την πλευρά του Συμβουλίου, σας υπόσχομαι ότι θα ασχοληθούμε με το ζήτημα αυτό, οδηγία δηλαδή για τους ναυτικούς, πάρα πολύ γρήγορα κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω και να σε ευχηθώ καλή εργασία. Η Ευρώπη μας διανύει σίγουρα μια δύσκολη περίοδο και βρισκόμαστε εμείς εδώ πέρα για να βρούμε λύσεις, ο καθένας στο πόστο του, ο καθένας στο ρόλο του, αλλά έχοντας ως συνεκτικό δεσμό τον ενθουσιασμό εκείνου που ξεκινάει μια περιπέτεια, μια καινούργια περιπέτεια για τη δημιουργία μιας καλύτερης Ευρώπης. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Αγαπητέ κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Μας δώσατε αρκετό υλικό ώστε να προχωρήσουμε σε διάλογο. Έχουμε εδώ τη λίστα, τον κατάλογο των ομιλητών. «22 συμπεριλαμβανομένων και των συντονιστών». Έχουμε χρόνο μέχρι τις 4.30 για να ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση. Αλλά να προτείνω το εξή. Στο πρώτο γύρο θα δώσω το λόγο στους συντονιστές των ε, κομμάτων, ανάλογα με το μέγεθος. Όμως θα σας παρακαλέσω να πάρετε το λόγο για δύο λεπτά Δεν πιστεύω ότι θα έχει κανείς πρόβλημα με αυτό και στο δεύτερο γύρο θα μπορέσουν να μιλήσουν οι υπόλοιποι που είναι στον κατάλογο των ομιλητών. Ο Ανδρέας τα έχει σημειώσει, όμως θα προτείνω να μην ε, ε, σπαταλήσουμε τον χρόνο και να βιαστούμε στο τέλος. ώστε άμα υπάρξουν, και, ε, ε, υπάρξει ενδιαφέρον και τελευταία στιγμή να μιλήσει κάποιο, να μπορέσουμε να δώσουμε το λόγο. Ξεκινάμε λοιπόν με τους συντονιστές. Και πρώτος θα μιλήσει ο συνάδελφος Μπέκα. Εκπροσωπώντας τον Ντάβιτ Κάζα που δεν είναι παρόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Μου αρέσει ο τρόπος που έχετε θέσει τις προτεραιότητες της Προεδρίας. Εστιάζεστε στην ανεργία. Και να γνωρίσω ότι η ανεργία των νέων είναι στην κορυφή των προτεραιοτήτων. Και αυτό έχει να κάνει με δύο θέματα που συζητήθηκαν υπό τις πέντε ε, προτεραιότητες, το πράσινη ανάπτυξη, η κοινωνική οικονομία. Να σας πω, να αναφερθώ εδώ σε αυτή τη στιγμή ε, πώς ενεργούν οι επιχειρήσεις, προσεκίζοντας, ε, έχοντας αυτή την προσέγγιση στην πράσινη, παράλληλα με την απασχόληση. Και στο θέμα της governance, να καλωσορίσω την έμφαση που έχει δώσει το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Υπάρχει περιθώριο ε, λύσεων και όσον αφορά τώρα την αδήλωτη εργασία θα μπορέσει να μας οδηγήσει σε πρόληψη, στην πρόληψη και στην πάταξη του φαινομένου αυτού. Και όσον αφορά την επέταξη του δικτύου για τις υπηρεσίες απασχόλησης, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην εκπαίδευση και στο ρόλο που παίζει και μιλάμε είτε για τυπική είτε για άτυπη εκπαίδευση και παράλληλα με την εμπλοκή των κοινωνικών εταίρων. Όλα αυτά τα θεωρώ πολύ σημαντικά. Θεωρώ ότι μπορούμε να μένουμε πολλά από την Ιταλική Προεδρία για την εύρεση Και εμείς από την πλευρά μας και ε, από την πλευρά του κόμματός μου σας διαβεβαιώ ότι θα υποστηρίξουμε αυτές τις πρωτοβουλίες σας. Ο λόγος στη Γιώτα Στάιντρουκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Με χαροποιεί ιδιαίτερα η πρόταση που κάνατε να συνεργαστείτε με το Κοινοβούλιο και τη συγκεκριμένη Επιτροπή. Γνωρίζετε ότι το Κοινοβούλιο χαίρεται πολύ όταν έχετε δυνατότητα να συνεργάζεται με το Συμβούλιο Επίσης, καλωσορίζω και τα σημεία έμφασης, όπως είναι ο διάλογος ε, για τη μακροοικονομική σταθεροποίηση. Θεωρώ ότι η Ευρώπη χρειάζεται ένα μηχανισμό για, ε, τον καιρό της κρίσης, χρειάζεται αλληλεγγύη, χρειάζεται ένα μηχανισμός αλληλεγγύης. Και φυσικά στη συνέχεια είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε αυτή τη συζήτηση επί της ουσίας. Όσον αφορά την καταπολέμηση της ενεργείας των νέων, θεωρώ ότι θα πρέπει το ταχύτερο δυνατό να προσπαθήσουμε να αφαρμόσουμε ε, αυτά που αποφασίσαμε ήδη. Την προηγούμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια του Στρασβουργού συζητήσαμε τις προθέσεις που έχουμε ως ε, Κοινοβούλιο. Αναφερθήκατε και στην κινητικότητα. Συμφωνώ με την εθελοντική κινητικότητα, αλλά και εδώ να δοθεί η έμφαση ότι η κινητικότητα από μόνη της δεν θα επιλύσει το πρόβλημα της νεανικής ανεργίας. Χρειαζόμαστε περισσότερα. Χρειαζόμαστε επενδύσεις για καλές θέσεις επασχόλησης. αφορά την ε, κοινωνική διάσταση της Νομισματικής Ένωσης. Επιτέλους χρειαζόμαστε και εκεί ε, πρόοδο ώστε τα κοινωνικά δικαιώματα να μην ε, υπολείπονται των οικονομικών ώστε να αποτρέψουμε το κοινωνικό ντάπινγκ και αυτό δεν αφορά μόνο ε, την αγορά και την ανάλυση της αγοράς αλλά θα πρέπει παράλληλα να θέσουμε δεσμευτικούς στόχους και να τους διερευνήσουμε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Τώρα για τους ναυτικούς είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι η ανταγωνιστικότητα δεν μπορεί να αποτελέσει τη μοναδική προσέγγιση. Στην Επιτροπή Απασχόλησης πρέπει από κοινού με εσάς να θέσουμε ε, σε πρώτη γραμμή ε, την ε, κατάσταση των εργαζομένων Ας περάσω τώρα στην πλατφόρμα για την ευήλωτη εργασία. Πρέπει και σε αυτό το θέμα να ε, διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει κοινό έλεγχος για αυτή την ε, πλατφόρμα και ότι θα υπάρχει ε, ε, ότι υπάρχει μια κοινή στάση, ότι δεν θα έχουμε 28 διαφορετικές μονόπλευρες στάσεις από τα κράτη-μέλη. Ευχαριστούμε, Γιώτα. Ο κύριος Μακεντάιρ από το ECR. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ κυρία Υπουργέ που ήρθατε εδώ για να μοιραστείτε μαζί μας τις σκέψεις σας κυρίως σχετικά με την ανάπτυξη και την απασχόληση. Θα έχετε πάρα πολύ φορτωμένο εξάμεινο σχετικά με το θέμα αυτό. Θα ήθελα να αναφερθώ σύντομα ε, στην ανεργία και απασχόληση των νέων, διότι είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτήν την Επιτροπή. Συνέχεια συζητούμε το θέμα αυτό. Είχαμε στο Στρασβούργο ένα ψήφισμα την περασμένη εβδομάδα και νομίζω ότι για να δημιουργήσουμε περισσότερες θέσεις εργασίας για τους νέους. Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον όπου οι επιχειρήσεις να μπορούν να αναπτυχθούν και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Ε, οι, Ευρω... Ε, οι Ευρωπαίοι Υπουργοί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορούν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, αλλά το κατάλληλο περιβάλλον και κυρίως οι μικρομεσές επιχειρήσεις, διότι οι περισσότερες, 85% των νέων θέσεων εργασίας προέρχονται από τις μικρομεσές. Πώς θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να δημιουργήσουν τις θέσεις αυτές. Ε, το θέμα το άλλο είναι ότι έχουμε επιχειρήσεις και εταιρείες ε, που χρειάζονται ε, που χρειάζονται νέους, αλλά οι νέοι που υπάρχουν δεν έχουν τα προσόντα. Θα πρέπει να υπάρχει μια αντιστοιχία. Τι έχετε να πείτε σχετικά με αυτό. Χαιρετίζω την ιδέα και διάβασα στο κείμενό σας του να μοιραστούμε τις βέλτιστες πραστικές. Νομίζω ότι στον τομέα της απασχόλησης υπάρχει ένα ρήγμα ανάμεσα στο βορρά και στο νότο. Δεν υπάρχει βεβαίως, δεν μπορούμε να πούμε ότι ένα μέγεθος ταιριάζει σε όλους, μια λύση είναι ιδανική για όλους. Αλλά θα ήθελα να δούμε, να ερευνήσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες τους τομείς όπου μπορούμε να έχουμε πολιτικές και πρακτικές που να λειτουργούν καλά και να μπορούν ε, να ανταλλαγούν, να μοιραστούν μεταξύ όλων. Και το τελευταίο ε, θέμα, ε, το, η ανάκτηση εργασιών από έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ξαναενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ήθελα τις απόψεις για το πώς θα μπορούσαμε να αυξήσουμε αυτήν την τάση επανόδου των θέσεων εργασίας ε, στην ε, Ευρώπη. Ε, Μαρία Νάρκιν, ε, εκ του Άλντε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ που ε, ήρθατε εδώ να μοιραστείτε τις σκέψεις σας μαζί μας. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να πω ότι η ομάδα μου θα υποστηρίξει τις προτεραιότητες σας. Έχω μερικές ερωτήσεις που θα ήθελα να σας θέσω. Μιλήσατε για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και την ανάγκη ε, να αυξήσουμε το συνέστημα του ανήκειν και θα ήθελα τις απόψεις σας για το πώς το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Διότι έχουμε την δημοκρατική νομιμότητα και αυτό χρειάζεται. Αναφέρατε την ανεργία των νέων ε, και τις μακροοικονομικές πολιτικές και πάλι Ξέρουμε περί τίνος πρόκειται, μιλήσατε για την ε, ποιότητα της εγγυήσεις της δημοσιονομικές. Υπήρξαν πρόοδοι, αλλά άνηση στα κράτη-μέλη. Το θέμα των πόρων δεν ξέρω αν είναι θέμα για τα κράτη-μέλη. Τις σκέψεις σας γι' αυτό μιλήσατε επίσης για την κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ και τους αυτόματους σταθεροποιητές. Το έχουμε συζητήσει το θέμα αυτό επανειλημμένα, μερικές φορές τουλάχιστον ε, στην Επιτροπή. Υπάρχει κάποια απτή πρόοδος που μπορείτε να μας αναφέρετε στο θέμα αυτό. Και ε, τελικά η κοινωνική οικονομία είπατε ότι ε, είναι ένα θέμα και μιλήσατε ε, για τη μόχλευση, για το θέμα της μόχλευσης. Έχετε κάποια πρωτοβουλία. Ίσως είναι κάτι που η Ιταλική ε, Προεδρία ε, ενδιαφέρεται για το θέμα αυτό και αν μπορούσατε να κάνατε κάποιες προτάσεις, να έχετε κάποια πρωτοβουλία σχετικά με την κοινωνική οικονομία, θα μπορούσε αυτό να παίξει σημαντικό ρόλο. Και νομίζω ότι είμαι ακριβώς στο χρόνο μου και λιγότερο από το χρόνο μου. Ήσουν όντως σύντομη. Τώρα στον κατάλογο έχουμε την Ροντιακάρη από την ΚΟΕ. Δεν είναι όμως παρούσα. Θα πάρει το λόγο αργότερα και ας περάσουμε στους πράσινους και στον Τζιν Λάμπερτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ την Ιταλική Προεδρία για την παρουσίαση. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που χαιρετίζομαι τουλάχιστον η ομάδα μου για την κοινωνική οικονομία για το βάρος της κοινωνικής διάστασης στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Θα ήθελα να ρωτήσω δύο πράγματα ε, σχετικά με το θέμα της καταπολέμησης της φτώχειας που αναφέρεται και αν ε, θα θέλατε όχι μόνο να αυξήσετε το εισόδημα από κάτω, αλλά να μειώσετε συνολικά τις ανισότητες μεταξύ των πτωχών και των πλουσίων και αν αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει τις συστάσεις για τους δείκτες ή τι θα μπορούσατε να προτείνετε για την αξιολόγηση των προτάσεων των κρατών μελών. Και σχετικά με τα όσα λέχθηκαν για την διακυβέρνηση και το θέμα του ανήκειν της ιδιοκτησίας, είναι η έλλειψη, έχουμε τη, στο, στην διαδικασία του εξαμήνου την έλλειψη της κοινωνίας των πολιτών, των εθνικών κοινοβουλίων σε πάρα πολλές χώρες, αλλά κάτι το οποίο νομίζω θα εξετάσετε εσείς. Και όσον αφορά στις ανισότητες, η Ιταλική Προεδρία ξέρω ότι προσπαθεί να δώσει ε, πνοή ε, σε, στην ε, νομοθεσία σχετικά με την οδηγία κατά των διακρίσεων. Μπορείτε να μας πείτε μερικά πράγματα για το θέμα αυτό. Και τελευταίο θέμα για από την άποψη της ομάδας μου σχετικά με την ανάπτυξη. Ε, μιλήσατε με τους Υπουργούς Οικονομικών για το θέμα των επενδύσεων ε, σχετικά με το θέμα των διεξιοτήτων, των προσόντων. Ίσως ε, αν έχουμε άτομα τα οποία είναι πάρα, που έχουμε πάρα πολλά προσόντα, αλλά δεν έχουμε επενδύσει ε, στον τομέα, τι γίνεται. Ευχαριστούμε. Από το EFD, ο επόμενος ομιλητής. Μινίστρο Καλησπέρα σας. Εδώ πέρα κάθομαι, κύριε Πολέτη, κύριε Υπουργέ. Αναφερθήκατε στη λεγόμενη κοινωνική κινητικότητα, ενώ στην Ιταλία μιλάμε περισσότερο για επισφαλείς θέσεις απασχόλησης, γιατί ξέρετε ότι υπάρχει κάτι το οποίο ονομάζεται ή ονομαζόταν κοινωνικό δίχτυ και το οποίο προστάτευε κατά κάποιο τρόπο τους πολίτες. Βλέπουμε όμως ότι η κινητικότητα πλέον αποτελεί υποχρέωση. Υποχρέωση πολλών ε, εργαζομένων οι οποίοι δεν έχουν άλλη εναλλακτική λύση και προκειμένου να διατηρήσουν μια θέση εργασία ανακάζονται να πάνε σε άλλε περιοχέ να μετεγκατασταθούν. Είναι υποχρεωμένοι να κάνουν κάτι τέτοιο. Η επισφαλή θέση απασχόληση λοιπόν θέση είναι ουσιαστικά μία πυλή, η ανασφάλεια αυτή είναι ουσιαστικά μία απειλή η οποία ουσιαστικά αφαιρεί από τους πολίτες, από τους εργαζομένους κάθε δυνατότητα, κάθε ικανότητα επενδύσεων όσον αφορά τον μέλλον τους. Ένας νέος ε, με επισφαλή θέση απασχόλησης παντρεύεται και θέλει να πάρει ένα στεγαστικό δάνειο, ξέρετε ποια είναι η απάντηση συνήθω τη τράπεζα. Αποκλείεται ποτέ ο άνθρωπο αυτό να πάρει δάνειο. Και να σα πω και κάτι ακόμα. Στον Ταβό, οι περισσότεροι οικονομολόγοι σε παγκόσμιο επίπεδο τόνισαν ότι ένα, το μεγαλύτερο ποσοστό του παγκόσμιου πλούτου βρίσκεται στα χέρια ελάχιστων ανθρώπων άνθρωποι που εκμεταλλεύονται τον πλούτο αυτό, εκμεταλλευόμενοι ουσιαστικά τους εργαζομένους παγκοσμίω. Διερωτάμε λοιπόν, μήπως θα έπρεπε να μην μιλάμε τόσο πολύ για αυτόματους σταθεροποιητέ, αλλά να μιλάμε περισσότερο για έναν ελάχιστο, αν μη τι άλλο, μισθό, για ένα επίδομα το οποίο θα μπορούσε να δίδεται σε όλους γιατί ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ο πλούτος, ο παγκόσμιος πλούτος να κατανέμεται ισότιμα σε όλους τους πολίτες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε με τους ε, συντονιστές, το από τη Κάρη, η οποία έχει φύγει από την αίθουσα. Φαντάζομαι ότι θα μπορέσουμε ε, να δώσουμε το λόγο αργότερα, κάποια στιγμή. 1,5 λεπτό από εδώ και πέρα ο χρόνος ομιλίας. Το θεωρώ ότι όμως είναι άδικο, πότε θα επιμείνω στα δύο λεπτά. Ας κάνουμε την πρώτη προσπάθεια με τον συνάδελφο Μπαχ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Υπουργό για την παρουσίασή σας. Έχετε ένα φιλόδοξο σχέδιο και σας εύχομαι καλή επιτυχία. Θα είμαι σύντομος για να εξοικονομήσω και χρόνο. Έχω δύο συγκεκριμένα ερωτήματα. Πρώτον, Κάνατε αναφορά στην πρωτοβουλία για την αδήλωτη εργασία και θεωρείτε ένα περαιτέρω πρόβλημα είναι το κοινωνικό dumping το οποίο το βλέπουμε και στις μεταφορές αλλά και σε άλλους ε, κλάδους, ε, στον κλάδο των ε, καθαριστών, καθαριστριών και των οικοδόμων. Θέλω να ρωτήσω αν θα το συζητήσετε το θέμα σε επίπεδο υπουργών και αν θα λάβετε μέτρα. Δεύτερον, αναφερθήκατε στην καταπολέμηση της φτώχειας και εδώ έχετε την υποστήριξή μου και θα ήθελα να σας ευχηθώ και καλή επιτυχία και να σας χαρώ αλλά μία παράκληση παράλληλα η πιο φτωχή από όλους είναι η άστεγη και θεωρώ ότι γίνεται πολύ λίγος λόγος για αυτούς. Επομένως, χρειάζεται και για αυτούς μία πρωτοβουλία Πολλές φορές σας ε, λέει η Επιτροπή ότι αυτό αφορά αρμοδιότητες ε, των κρατών μελών, όμως θα ήθελα να σας παρακαλέσω να ξεκινήσετε και σε αυτό το τομέα μια πρωτοβουλία. Ευχαριστώ πολύ. Η Ελένη Τζεντήλε στη συνέχεια. Καλημέρα σας Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε Υπουργέ Πολέτη. Άκουσα με ιδιαίτερα ενδιαφέρον ε, την παρέμβασή σας και συμφωνώ με ορισμένα από τα πράγματα τα οποία είπατε όσον αφορά τις προγραμματικές δηλώσεις της Ιταλικής Προεδρίας. Θα ήθελα όμως να προσθέσω και κάποια ακόμα στοιχεία προκειμένου να κάνουμε και μία συζήτηση η οποία θα λαμβάνει υπόψη της και κάποιες άλλες πτυχές και κάποια άλλα θέματα τα οποία δεν θα πρέπει να παραβλέπουμε. Πρώτον, η εργασία και απασχόληση των γυναικών, καθώς επίσης και το ζήτημα της συμφιλίωσης προσωπικής και επαγγελματική ζωής. Επομένως, να δούμε τελικά ποιες είναι οι πολιτικές εκείνες οι οποίες έχουν στο κέντρο τους τα δικαιώματα αυτά των γυναικών και κυρίως το δικαίωμα συμφιλίωσης επαγγελματικής ε, προσωπικής ζωής. Πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν λοιπόν οι γυναίκες επαγγελματικές προκλήσεις διατηρώντας παράλληλα την προσωπική του ε, ζωή. Ξέρετε επίσης ότι υπάρχουν πάρα πολλοί και πάρα πολλές γυναίκες οι οποίες αποκλείονται, εκδιώχνονται θα έλεγα, από την αγορά εργασίας. Νομίζω ότι θα πρέπει να αξιολογήσουμε πολύ πιο προσεκτικά το ζήτημα αυτό και να δούμε επίσης συγκεκριμένα πώς η εγγύηση αυτή για τους νέους, την οποία αναφέρουμε τόσο συχνά, μπορεί τελικά να εφαρμοστεί στην πράξη και να δούμε για παράδειγμα τι γίνεται σε ορισμένες περιοχές όπως τη δική μου την περιφέρεια. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει να έχουμε κατά νου και κάποια άλλα συστήματα, κάποιους άλλους τομείς, για παράδειγμα τους εργαζόμενους εκείνους οι οποίοι αποκλείονται από την αγορά εργασίας για τον έναν τον άλλο χώρο ή εκδιώχνονται από κάποιες επιχειρήσεις και να ασχοληθούμε προφανώς και με το ζήτημα της αδήλωτης εργασίας. Κύριε Υπουργέ, λοιπόν, νομίζω ότι στα πλαίσια της συζήτησης που θα κάνουμε και στα πλαίσια της συνεργασίας που θα έχουμε, θα πρέπει οι προτάσεις μας να είναι καθαρά οριζόντιες και να λαμβάνουν υπόψη τους ζητήματα τα οποία απασχολούν και άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές. Για παράδειγμα, το ζήτημα της μετανάστευσης είναι ένα ζήτημα οριζόντιο, το οποίο ουσιαστικά επηρεάζει και τις δικές σας πολιτικές και τις δικές σας αρμοδιότητες και πλήττει πάρα πολύ κάποιες χώρες όπως η Ιταλία, η οποία σε καθημερινή βάση καλείται να αντιμετωπίσει το ζήτημα αυτό, το οποίο συμβάλλει προφανώς και στην φτώχεια ή την υπερβολική θα έλεγα μάλιστα φτώχεια. Νομίζω λοιπόν ότι ε, μπορούμε αυτή τη στιγμή να ξεκινήσουμε μια σημαντική εργασία βασιζόμενη στην πολύ καλή εμπειρία την οποία έχουμε, έχοντας βέβαια και την δική σας τη συμμετοχή και τη συμμετοχή των συναδέλφων σας ε, στην κυβέρνηση για τα ζητήματα βέβαια που άπτονται την αρμοδιοτήτων τους. Καλή εργασία κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ. Ο στον Τόμας Μαν. Ευχαριστώ. Είπατε ότι η πρώτη προτεραιότητα είναι η καταπολέμηση της ενεργείας των νέων. τελευταία φορά, στην, ε, τελευταίο χρόνο στην Επιτροπή προσπαθήσαμε να ε, έχουμε μια πρόταση για μια εγγύηση νέων. Είναι κάτι πολύ φιλόδοξο αυτό, ως διατύπωση αυτή η εγγύηση. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ασχοληθούμε σοβαρά με αυτό το θέμα και να πω κάποια πράγματα ακόμα. Το θέμα είναι πώς θα το εφαρμόσουμε. Τα 6 δισεκατομμύρια που έχουμε είναι λίγα σε πρώτη φάση, όμως είναι μια αρχή. Πώς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό κύριε Υπουργέ. Από τον Ιανουάριο του φετινού έτους υπάρχουν αυτά τα χρήματα, αλλά υπάρχουν κράτη που δεν τα έχουν λάβει ακόμα. Πρέπει να αιτιολογήσουν για ποιο λόγο θέλουν να τα λάβουν και να το αιτιολογήσουν. Όμως είναι όλα, περιμένει μέχρι οι αρμόδιες αρχές να είναι σε θέση να ε, κάνουν αυτό που πρέπει. Πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό και αυτό πρέπει να το κάνετε ε, εσείς. Έθεσα μια ερώτηση και περιμένω απάντηση. Είμαι και σε μια άλλη επιτροπή και η απάντηση θα, ε, γίνει, θα την ακούσετε και εσείς. Ελπίζω να μπορέσετε να κάνετε κάτι και για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ, Τόμα. Πράντο Μπενεφίτσι στη συνέχεια. Μπενιφέι, με συγχωρείτε, λέει ο πρόεδρο. Υπάρχουν διαφορέ ανάμεσα σε προφορές, λέει ο Πρόεδρο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ και παίρνω τον λόγο ως μέλος της κοινοβουλευτικής αυτής Επιτροπής Απασχόλησης Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο Γιούνκερ στην προηγούμενη σύνοδο Ολομελίας πήρε το λόγο και αναφέρθηκε με απόλυτη σαφήνεια στο ότι θα πρέπει η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ασχοληθεί όλος ιδιαίτερος με την καταπολέμηση της ανεργίας και ιδιαίτερα για την καταπολέμηση ανεργίας των νέων. Εμείς εγκρίναμε ένα ψήφισμα ίδιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην προηγούμενη σύνοδο και στο ψήφισμα αυτό θέτουμε συγκεκριμένα ζητήματα. Αναφερθήκαμε συγκεκριμένα στο ζήτημα της διακριτικής μεταχείρισης όσον αφορά τους νέους από διάφορες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είδαμε για παράδειγμα ότι υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα ανεργία σε διαφορετικές χώρες προφανώς και είπαμε επίσης ότι θα πρέπει να ενισχυθεί περισσότερο η κινητικότητα των νέων όσον αφορά τις αγορές εργασίας προκειμένου να καταφέρουμε να ενισχύσουμε περισσότερο και την ενιαία αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω λοιπόν ότι είναι απαραίτητο να καταβληθούν οι απαραίτητες προσπάθειες, οι οποίες έχουν ήδη ξεκινήσει κάποιες κυβερνήσεις όπως η Ιταλική, προκειμένου να καταφέρουμε να αυξήσουμε κάπως τις ποσοστώσεις, όπως για παράδειγμα ποσοστώσεις συγχρηματοδότησης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, προκειμένου να απελευθερωθούν περισσότερα κονδύλια κοινοτικά σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, για να αυξηθούν οι πόροι εκείνοι τελικά, οι οποίοι δίνονται, χρησιμοποιούνται για νέες θέσεις απασχόλησης. Εν κατακλείδη δύο συγκεκριμένα αιτήματα, κύριε Υπουργέ. Πρώτον, σε σχέση με τα όσα έχουν υποθεί μέχρι στιγμή. Μπορείτε να μα πείτε περισσότερα και πιο συγκεκριμένα πράγματα όσον αφορά την ανάπτυξη του δικτύου Έουρε. Πολλέ φορέ το αναφέρατε αυτό στο λόγο σα. Και αναφέρομαι σε αυτό γιατί το ζήτημα των υπηρεσιών απασχόληση και εργασία είναι υπηρεσίε πολύ σημαντικέ για τι χώρε μα. Οι υπηρεσίε αυτέ πολλέ φορέ δεν είναι το ίδιο αποτελεσματικέ από τη μία χώρα στην άλλη. Δεύτερον, ένα ζήτημα το οποίο θέσαμε και στα πλαίσια του ψηφίσματός μας την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά και ως Ιταλοί ευρωβουλευτές στις επαφές που είχαμε με τον Υφυπουργό Γκότσι, το ζήτημα των αυτόματων σταθεροποιητών. Πώς προχωράει το ζήτημα αυτό, σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε, γιατί θεωρώ ότι είναι μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες της Ιταλικής Προεδρίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να σας υπενθυμίσω το περιθώριο των δύο λεπτών. Ε, ο λόγος στη Βερόνικα Λούπε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Υπουργέ που ήρθατε εδώ, εδώ σε αυτήν την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής μας αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό το οποίο που σας ακούσαμε εδώ να παρουσιάζετε τις προτεραιότητες της Προεδρίας σας. Θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή τύχη. Είναι σημαντικό ε, για όλες τις χώρες ε, να τηρηθούν αυτές οι προτεραιότητες και να εκπληρωθούν αυτοί οι στόχοι. Πολλοί αναφέρθηκαν στα θέματα αυτά πριν από μένα, δεν θα ήθελα να τα επαναλάβω, θα επιμείνω πάνω στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Στην προηγούμενη θητεία είχαμε μια συμφωνία για τα διάφορα στοιχεία. Θα ήμασταν ευτυχείς αν μπορούσαμε να συζητήσουμε πριν από το Συμβούλιο όλα αυτά τα στοιχεία. Η στρατηγική 2020 είναι βεβαίως σημαντική για την καταπολέμηση της ανεργίας, αλλά πρέπει να δούμε ίσως να, θα έπρεπε ίσως να αναθεωρήσουμε τις φιλοδοξίες σε σχέση με το τι είναι φυκτό. Κάτι άλλο είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει καλύτερος συντονισμός ανάμεσα στις δημόσιες υπηρεσίες που ασχολούνται με την απασχόληση. Όντως, Ορισμένοι τόνισαν τον υποχρεωτικό χαρακτήρα, άλλοι πιστεύουν ότι θα πρέπει να γίνεται αυτό σε εκούσια βάση. Ας μιλήσουμε τώρα για την εγγύηση για τους νέους. Από πού θα προέλθουν τα νέα κονδύλια. Θα αυξηθεί ο προϋπολογισμός που προβλέπεται για αυτήν την πρωτοβουλία για τους νέους από το 16. Ε, ξεπερνάω βεβαίως τα δύο λεπτά, τώρα εδώ. Μιλήσατε και για διακρίσεις, δεν πρέπει να μιλήσουμε και για τους Ρωμά. Υπάρχει ε, κάποια η πρωτοβουλία για αυτόν τον πληθυσμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ Μαρίτα Ουσκο. Ευχαριστώ κύριε Πολέτη. Δεν έχω μετάφραση στα σουηδικά. Θα προσπαθήσω να μιλήσω με τα αγγλικά που γνωρίζω. Φιλόδοξο το πρόγραμμά σας και πολύ καλό αυτό της Θελικής Προεδρίας. Τα έχετε συμπεριλάβει όλα στην ατζέντα σας. Παρόλο που είναι πολύ σημαντικό να μην ξεχνάμε να μην ξεχνάμε το πρόβλημα που οδηγεί σε εξτρεμιστικές τάσεις σε όλη την Ευρώπη. Κάποιοι είναι απελπισμένοι να βρουν εργασία και κάποιοι εργοδότες το χρησιμοποιούν αυτό για να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον ανασφάλειας με χαμηλά, χαμηλές αμοιβέ, με αδήλωτη εργασία με επισφαλείς συνθήκες εργασίας και αυτό είναι κάτι ιδιαίτερα επικίνδυνο στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Οπότε μας ικανοποιεί η εστίαση που δίνεται στην κοινωνική διάθεση και στην οικονομική πολιτική, στην ανεργία των νέων. Όμως παράλληλα είναι πολύ σημαντικό να φροντίσουμε ώστε να υπάρχουν δίκες αμοιβέ. Και αυτό είναι από τα κεντρικά θέματα που θα ήθελα να προσθεθεί στην ατζέντα σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πολέτη. Στην Τανούτα Γεζοβιέτσκα περνάμε τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ την Ιταλική Προεδρία που έχει μεταξύ των προτεραιοτήτων της σημαντικά θέματα για αυτήν την Επιτροπή. Μια από τις προτεραιότητες είναι να προωθηθεί η απασχόληση των νέων και από το 2013 ε, δύο εκατομμύρια θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν στην Ευρώπη που είναι ακόμα κενές αυτές οι θέσεις εργασίας, διότι δεν υπάρχει αντιστοιχία ανάμεσα στα προσόντα που ζητούνται και στην προσφορά των προσόντων. Θα ήθελα να μου πείτε τι σκέπτεστε γι' αυτό, τι θα κάνετε. Ο Τόμας Μαν είπε ότι θα πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί. Θα ήθελα να δω πόσο αποφασιστική θα είναι η Ιταλική Προεδρία Χαίρομαι που μια από τις προτεραιότητες σας είναι η υποστήριξη των κοινωνικών επενδύσεων στην Ευρώπη για να βελτιωθεί η ποιότητα και σταθερότητα των κοινωνικών μοντέλων. Το Νοέμβριο 2012 υιοθετήθηκε η έκθεσή μου για τις κοινωνικές επενδύσεις όπου κάναμε έκκληση στα κράτη-μέλη να αναθεωρήσουν τα κοινωνικά τους ε, συστήματα και από το κράτος πρόνοια να προχωρήσουν προς ένα κράτος όπου οι πολίτες θα είναι πιο δυναμικοί, πιο ενεργητικοί. Πώς η Προεδρία θα ασχοληθεί με μια πραγματική μεταρρύθμιση του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Και ένα τελευταίο πράγμα είναι η προσπάθεια για ε, τήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Ποιες είναι οι πιθανότητες να δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, της εργασίας που δεν υπόκειται σε κανονισμούς αν η Ιταλική Προεδρία αλλά κάνει ένα βήμα, έστω λάβει και ένα μέτρο για τις προτεραιότητες που αναφέρεται, θα έχουμε μεγάλη επιτυχία, διότι ένα βήμα είναι καλύτερο από πολλά μικρά βήματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ζήων Σίμων στη συνέχεια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον Υπουργό. βάζετε την ανεργία των νέων στο επίκεντρο των ε, θεμάτων σας και είπατε στην ε, σελίδα 44 ε, του αγγλικού κειμένου που αναφέρεται η ρίστο εμπαρόδο στα μέτρα για την καταπολέμηση της υπερβολικής επισφάλειας. Θα ήθελα να σχολιάσω και να πω αν υπάρχει κίνδυνος ίσως να εστιαστούμε πολύ περισσότερο στα μακροοικονομικά, στην ποσότητα των θέσεων εργασίας, εις βάρος της ποιότητας τους. Ένας νέος στην περιφέρειά μου χτες μου είπε ότι οι συνάδελφοί του εργάζονται σε βάρδιες 27 ωρών στο Μακδόναλντ αποτελεσματικά. Να έχουμε μισό εκατομμύρια νέους σε θέσεις εργασίας στο Μακδόναλντ με βάρδιες 27 ωρών. Θα έχουμε κάνει ένα καλό πράγμα. Δεν νομίζω. Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε ένα τέσσερα ε, εκατομμύρια άνθρωποι με ε, συμβόλαια μηδενικά, με ε, προσωρινά αυτοαπασχολούμενος. Το θέμα της επισφάλειας νομίζω ότι είναι ένα σοβαρό πρόβλημα σχετικά με την ποιότητα της εργασίας. Και θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για τα μέσα με τα οποία η Ιταλική Προεδρία θα μπορούσε να προωθήσει την ποιότητα και όχι μόνο την ποσότητα, τον αριθμό, διότι οι νέοι περισσότερο από τους άλλους υποφέρουν από, αυτήν, από την έλλειψη ποιότητας στην αγορά εργασίας. Ευχαριστώ. Ο Άρνε Γκέρικε έχει το λόγο. Είναι εκτός μικροφώνου ο μιλητής. Εκτός μικροφώνου ο μιλητής. Λοιπόν, να ξανασπαθήσω. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ, κύριε Πολέτη. Είναι στόχος της τελικής Προεδρίας να θέσει στόχους για μια Ευρώπη φιλική προς τα παιδιά. Θεωρείτε την ίδρυση μιας πλατφόρμας για την οικογένεια κατάλληλη για να προσαρμοστεί η ευρωπαϊκή πολιτική γιατί στο θέμα της ενεργείας των νέων πιστεύω ότι πρέπει να ε, προληπτικά μέτρα. Θεωρώ ότι η βελτίωση της οικογενικής πολιτικής έχει σχέση με αυτό και με ένα τέτοιο τρόπο να γίνει αυτό, ώστε να είναι ε, η προσπάθεια βιώσιμη. Ελπίζω η Ιταλία να παίξει ε, πρωτοποριακό ρόλο σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος στην Ουλρίκε Τρεμπέζιους. Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσω που μας παρουσιάσατε το πρόγραμμά σας σήμερα και όταν κάνετε λόγο για ανεργία των νέων τότε σίγουρα ένα από τα πιο σημαντικά θέματα είναι η επένδυση στην διαβίω εκπαίδευση. Θα ήθελα να ξέρω τι ακριβώς εννοείται ως προς τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την καταπολέμηση της ενεργεια των νέων. Έχοντας κατά νου ότι η αιτία για αυτή την ανεργία θα πρέπει να διερευνηθεί αλλά να ληφθεί υπόψη ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ε, προσφέρουν θέσεις εργασίες για τους νέους, κυρίως μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν υπόκεινται σε υπερρύθμιση και έχει περιοριστεί η ανταγωνιστικότητά τους. Θα ήθελα να μάθω τι μπορεί να γίνει σε αυτό το θέμα μελλοντικό για να αποτραπεί αυτή η υπερρύθμιση και αυτό που μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον είναι η αναφορά που κάνατε ότι στις πρώτες διαπραγματεύσεις στο Μιλάνο ότι εκεί συζητήθηκε ένα κοινό κοινωνικό ε, σύστημα, ένα κοινωνικό σύστημα ασφάλισης. Θα ήθελα να ξέρω ακριβώς τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτό το σύστημα και το οποίο συζητήσατε. Ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος του Richard Uh, uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να σας μιλήσω για την ε, κοινωνική ευθύνη. Ε, είμαι και εισηγητής και ξέρω ότι το Υπουργείο σας είναι υπεύθυνο με άλλο Υπουργείο και λέτε ότι έχετε θα κάνετε διάφορες παρεμβάσεις τι ε, προγραμματίζεται. Επίσης, η γνώμη για την οδηγία σχετικά ε, με τις μη οικονομικές αναφορές και που συμφωνήθηκε επί ελληνικές προεδρίας. Ε, πότε θα επιβεβαιωθεί στο Συμβούλιο αυτή η συμφωνία και πώς θα προχωρήσετε σε σχέση ε, με την ε, κοινωνική ευθύνη και την ευθύνη αποζημιώσεων ε, και και επίσης στο Συμβούλιο για την Αϊφόρο Ανάπτυξη πρόκειται να, αυτό που σας προτείνετε να το δεχτείτε. Επίσης, εσείς και η κυβέρνησή σας θα πρέπει σε συνολικό επίπεδο να εφαρμόσετε τα κατευθυντήριες γραμμές των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα ε, της εργασίας. Όλα τα κράτη-μέλη έχουν κληθεί να υποβάλουν προγράμματα δράσης. Θα χρησιμοποιήσετε την Προεδρία σας όχι μόνο για το δικό σας πρόγραμμα δράσης, αλλά για να ενθαρρύνετε άλλα κράτη να το πράξουν. Ευχαριστώ. Λόγος στην κυρία Μέρα Μπιτσότο. Καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που μιλάμε πάρα πολύ για απασχόληση και εργασία αλλά στην πράξη κάνουμε ελάχιστα πράγματα. Και εσείς ουσιαστικά συνεχίζετε την παράδοση αυτή, ωραία λόγια, λίγες πράξεις όμως. Η Ευρωπαϊκή Ένωση απαρτίζεται από 28 κράτη-μέλη, 28 λοιπόν διαφορετικές οικονομίες, 28, 28 διαφορετικά εργατικά δίκαια, 28 διαφορετικά φορολογικά συστήματα. Βλέπετε για παράδειγμα πόσο διαφέρει η Ιταλία από κάποιες άλλες χώρες. Μιλάμε όμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενία αγορά έχοντας εντελώς διαφορετική τελικά κατακαιρματισμένη βάση από χώρα σε χώρα. Εσείς τι θα κάνετε για να αρμονίσετε τους κανόνες αυτούς γιατί αν δεν το κάνετε αυτό θα έχουμε πάντα κανόνες ε, κατηγορίας Α, συγγνώμη χώρες που θα ανήκουν στην κατηγορία Α και χώρες οι οποίες θα ανήκουν στην κατηγορία Β, σε υποδιέστερη δηλαδή θέση. Επίσης, ας μην ξεχνάμε ότι ένας τεράστιος αριθμός ανέργων βρίσκεται στην Ιταλία, εξίσου πάρα πολλοί άνεργοι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα επίσης να πείτε στον κύριο Αλφάνο, τον Υπουργό Εσωτερικών, ότι δεν χρειαζόμαστε περισσότερους μετανάστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας βοηθήσουμε τους μετανάστες στη χώρα τους. Δεν μπορούμε να φέρνουμε στην Ιταλία περισσότερους ανθρώπους οι οποίοι δεν πρόκειται ποτέ να βρουν καμία θέση απασχόλησης. Ο κύριος Γιούνκερ πριν από μερικές μέρες βέβαια μας είπε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα επόμενα χρόνια θα έρθουν 50 εκατομμύρια νέοι μετανάστες. Φαίνεται να συμφωνεί πάντως και ο κύριος Γιούνκερ με τον κύριο Αλφάνο. Ευχαριστώ πολύ Γεώργη Πυρίσκη, ο επόμενος ομιλητής. Κύριε Υπουργέ, στις γραπτές προτεραιότητες της Ιταλικής Προεδρίας αναφέρεται ότι η οικονομική κρίση απέδειξε, εδώ είμαι, εδώ βρίσκομαι, απέδειξε ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις πρέπει να συνοδεύονται με μέτρα που να εξασφαλίζουν κοινωνική συνοχή. Πιστεύετε ότι η έννοια της κοινωνικής συνοχής θα μπορεί να είναι στο επίκεντρο της συζήτησης για τις κοινωνικές πολιτικές και κοινωνική διάσταση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, διότι από τις ερωτήσεις που ακούσατε μέχρι τώρα καθίσταται σαφές ότι υπάρχει μια ολόκληρη σειρά επιγόντων προβλημάτων που σχετίζονται με την κοινωνική συνοχή και υπάρχουν και προκλήσεις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες. Σε αυτό το κοινοβούλιο έχουμε να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση του να καταστήσουμε την Επιτροπή αυτή πάρα πολύ δυναμική, ε, πολύ προοδευτική. Ε, ποιος θα είναι ο διάλογός σας σχετικά ε, με το θέμα αυτό, με τον Υπουργό Παντοβά. Ευχαριστώ, Κριστίνα Μορβάη, στη συνέχεια. Köszönöm miniszter úr, magyar képviselőként olyan kérdéseket Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ως Ευρωβουλευτής από την Ουγγαρία θα ήθελα και εγώ να θέσω με τη σειρά μου κάποια ερωτήματα, ιδίως όσον αφορά τις προτεραιότητες της Ιταλικής Προεδρίας. Τα ερωτήματά μου έχουν να κάνουν κυρίως με τα κράτη-μέλη εκείνα τα οποία θεωρούνται λίγο κράτη-μέλη δεύτερης κατηγορίας. Μια βασική όμως προτεραιότητά μας θα πρέπει να είναι προφανώς, όπως το είπατε και εσείς, η ανεργία των νέων. Υπάρχουν ε, πολλοί νέοι στη χώρα μου, την Ουγγαρία, οι οποίοι αναγκάζονται να πάνε σε άλλες χώρες για να βρουν μια θέση απασχόλησης. Ουσιαστικά πρόκειται για πραγματικούς οικονομικούς πρόσφυγες. Πολύ συχνά επίσης εργάζονται σε άθλιες συνθήκες στις άλλες χώρες και αναγκάζονται προφανώς να ξεριζωστούν από τη χώρα τους εγκαταλείποντας οικογένεια, παιδιά, συζύγους κτλ. Είναι φυσιολογικό αυτό το πράγμα. Είμαι νέα στην Επιτροπή αυτή, αλλά πώ άκουσα η Επιτροπή Απασχόλης και Κοινωνικών Υποθέσεων τελικά αποδέχεται την κατάσταση αυτή ως φυσιολογική. Εγώ θεωρώ ότι σημαίνει ακριβώς το αντίθετο. Πρέπει να αλλάξει η πρακτική αυτή. Τώρα όσον αφορά τη φτώχεια, την ένδεια. Γνωρίζετε κύριε Υπουργέ ότι στην Ουγγαρία υπάρχουν ορισμένοι εργαζόμενοι οι οποίοι κάνουν πολύ επίπονη σωματική εργασία για 8 ώρες την ημέρα έχοντας μόνο 200 ευρώ μισθό το μήνα σε εργοστάσια μάλιστα που ανήκουν σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, σε επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ίδιες αυτές επιχειρήσεις, οι στιγατρικές που έχουν στην Δυτική Ευρώπη πληρώνουν 5, 6, ακόμα και 7 φορές το μισθό που δίνουν στους εργαζομένους στην Ανατολική Ευρώπη. Είναι φυσιολογικό αυτό το πράγμα, πιστεύετε ότι κάτι πρέπει να κάνουμε για να πατάξουμε και το φαινόμενο αυτό. Για παράδειγμα, αν μη τι άλλο, να υποχρεώσουμε τις επιχειρήσεις αυτές να δίνουν έναν ελάχιστο μισθό, να μην μπορούν να κατεβούν κάτω από ένα συγκεκριμένο κατόφλι όσον αφορά το μισθολογιό τους. Τρίτον, η TTIP, e η Συμφωνία Εμπορικών Συναλλαγών και Επενδύσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών, Πώς θα επηρεάσει, πιστεύετε, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς θα επηρεάσει τους ίδιους εργαζομένους. Όταν θα συζητήσουμε για τη συμφωνία αυτή, την TTIP, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην εκπροσωπηθεί εδώ πέρα με αξιωματούχους μόνο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και με εκπροσώπους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, να μας πούνε και αυτή την άποψή τους. Ευχαριστώ, Σίλβιο Κώστα. Η κυρία Σιλβία έχει το λόγο. στον κύριο Λάμπρο Φουντούλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ε, αξιότιμε κύριε Υπουργέ. Όσον αφορά την αδήλωτη εργασία, δεν είναι μόνο η σφοροδιαφυγή και η φοροδιαφυγή που έχουν επίπτωση στις οικονομίες των χωρών. Υπάρχουν επιπτώσεις στην υγεία, από την αδίλωτη εργασία ατόμων συνήθως παράνομων μεταναστών που γίνονται θύματα εκμετάλλευσης των εργοδοτών. Υπάρχει κίνδυνος δημόσιας υγείας όταν τα άτομα αυτά δεν έχουν περάσει από υγειονομικό έλεγχο και απασχολούνται σε καταστήματα συνήθως παρασκευαστήρια, υγειονομικού ενδιαφέροντος, κουζίνες, εστιατορίων κλπ. Είναι πολύ εύκολος ο τρόπος αντιμετώπισης της αδίλωτης εργασίας. Εάν σταματήσει η πληρωμή των εργαζομένων με μετρητά, και πληρώνονται μέσω τράπεζας με κάρτα μισθοδοσίας. Κανένας εργοδότης να μην μπορεί να δικαιολογήσει έξοδα μισθοδοσίας για απασχόληση εργαζομένων εάν αυτοί δεν πληρώνονται μέσω τράπεζας. Θα πρέπει να παρακρατούνται οι ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές εισφορές αυτόματα ώστε να αποφεύγεται η φοροδιαφυγή και η εισφοροδιαφυγή. Αυτό θα είναι ένας τρόπος να αποτρέπεται η παράνομη μετανάστευση από άτομα που θεωρούν ότι θα επιβιώσουν στις συνθήκε όπου υπάρχει κρατική ολιγορία στο θέμα ελέγχου των συνθήκων εργασία. Αυστηρέ ποινέ, κυρίω σε εργοδότε προσπαθούν να εκμεταλλευτούν του εργαζόμενου λόγω κρίση, προσφέροντα δουλειά με χαμηλό μισθό και χωρί ασφάλεια. Να μην αποκλείεται κανεί από την αγορά εργασία, παρά μόνο οι παράνομοι μετανάστε, οι οποίοι εύκολα θύματα των εργαδοτών στερούν θέσει εργασία από του πολίτε τη χώρα. Ειδικά σε χώρε με υψηλά ποσοστά ανεργία και ειδικότερα στου νέου, το φαινόμενο έχει πάρει εκρηκτικέ διαστάσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει με την πλατφόρμα και με τη συνεργασία των κρατών μελών και φορέων να δώσει κατευθυντήριε γραμμέ για την εξάλληψη του φαινομένου. Για του μετανάστε, οι οποίοι έχουν έρθει παράνομα στη χώρα, θα πρέπει οι κυβερνήσει να μεριμνήσουν για την ανθρώπινη διαβίωσή του μέχρι να επαναπατριστούν στι χώρε καταγωγή του. Εάν περιμένουμε από τι υπηρεσίε των χωρών, δηλαδή επιθεωρήσει εργασία, υπηρεσίε κοινωνική ασφάλεια, φορολογικέ αρχέ κτλ. για την αποτροπή τη αδήλωτης εργασία, θα, το είχα, θα είναι ένα θέμα που θα το είχαν κάνει χρόνια τώρα. Αντί να πατάξουν την εσφοροδιαφυγή ώστε να μην έχουν πρόβλημα τα ταμεία, μειώνουν τι συντάξει από ανθρώπου που δούλευαν για μια ζωή, περιμένοντα τα γεράματά του να μπορούν να ζουν αξιοπρεπώ. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εδώ κλείνει ο κατάλογος των ομιλητών. Κύριε Υπουργό, ε, κύριε Υπουργέ, είχαμε μια ζωντανή συζήτηση. Ελπίζω να μην ήταν πολλά αυτά που υποσχεθήκα. Δεν θα ήταν τόσο χρονικό περιθώριο. 22 ερωτήσεις σας τέθηκαν. Ο λόγος σας κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω όλους για τις ευχές σας καταρχάς, για τις ερωτήσεις και τις παρατηρήσεις σας. Στην ουσία είναι πάρα πολύ δύσκολο να απαντήσω ξεχωριστά σε κάθε ερώτηση, ωστόσο θα προσπαθήσω στην απάντησή μου να εντάξω στο δυνατόν περισσότερα ερωτήματα και βέβαια θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος και αναγκαστικά η απάντησή μου θα είναι και κάπως γενική. Ωστόσο θα προσπαθήσω όπως σας πέν εντάξω τα περισσότερα ερωτήματα στην απάντηση αυτή. Μια πρώτη ερώτηση και μια πρώτη απάντηση. Όσον αφορά τις φιλοδοξίες της Ιταλικής Προεδρίας, όσον αφορά τις βασικέ προτεραιότητες και το εξάμεινο. Εγώ θεωρώ πραγματικά ότι ε, συντοποιούμε όλοι ότι κατά τη διάρκεια του εξαμήνου αυτού ο χρόνος είναι τελικά ελάχιστος, είναι πάρα πολύ σύντομος. Πρέπει να περιμένουμε και τη σύσταση της Νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξέρουμε πάντως ότι πρόκειται για το πρώτο εξάμεινο μιας νέας νομοθετικής περίοδου. Επομένως οι συζητήσεις που θα κάνουμε κατά τη διάρκεια του εξαμήνου αυτού, τα επιχειρήματα τα οποία θα καταφέρουμε να ανταλλάξουμε, τα ζητήματα που θα θέσουμε στο προσκήνιο είναι ζητήματα τα οποία προφανώς θα ξεπεράσουν το Ιταλικό που θα απασχολήσουν προφανώς και τις επόμενες ε, προεδρίες. Επομένως ε, γνωρίζουμε τα βασικά όρια, τους περιορισμούς που υπάρχουν στα πλαίσια της Ιταλικής Προεδρίας, τους χρονικούς περιορισμούς. Ξέρουμε όμως ότι αν έχουμε την καλύτερη δυνατή συνεργασία μεταξύ Κοινοβουλίου, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Συμβουλίου, τότε οι πρωτοβουλίες αυτές μπορούν πραγματικά να πάρουν μια πιο μακροπρόθεσμη διάσταση και να θέσουμε τελικά επιτάπητος κάποια ζητήματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά όχι μόνο για το επόμενο εξάμεινο αλλά γενικότερα για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μας είπατε, ρωτήσατε πάρα πολύ τι μπορεί να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν μη τι άλλο αυτή τη στιγμή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να δώσει ένα προσανατολισμό, να στείλει ένα μήνυμα, να πει τι ακριβώς θέλει, τι θα ήθελε να πετύχει, ποιες είναι οι επιθυμίες, ποιες είναι οι προσδοκίες του. Μπορεί να πιέσει προκειμένου τα πράγματα τελικά να πάρουν μια συγκεκριμένη ρότα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ακολουθήσει ενδεχομένω το δικό τη δρόμο, το Συμβούλιο το δικό του, αλλά αν μη τι άλλο μπορούμε εξ αρχή να έχουμε ένα συντονισμένο παραγωγικό διάλογο. Αν το πετύχουμε αυτό από μόνο του, αυτό αποτελεί ένα σημαντικότατο επίτευγμα. Να δώσω τώρα κάποιες απαντήσεις όσον αφορά το ζήτημα του εξαμήνου, του σχετικού σχεδίου δηλαδή. Εν γέννη, εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε έναν πιο επικοδομητικό διάλογο σε θεσμικό επίπεδο, προκειμένου να καταφέρουμε να έχουμε έναν μόνιμο τέτοιο διάλογο και τα επόμενα χρόνια και συντοποιούμε επίσης ότι θα πρέπει πολλές φορές να κάνουμε ένα διάλογο όχι μόνο μεταξύ θεσμικών οργάνων, αλλά και μεταξύ διαφορετικών επιμέρους οργάνων αυτών των θεσμικών οργάνων, για παράδειγμα ομάδες εργασίας του Συμβουλίου. Θα γίνει πάντως μια συζήτηση μεταξύ Υπουργών Εκπαίδευσης και Υπουργών Εργασίας. Ξεκινήσαμε την όλη συζήτηση για το ζήτημα των αυτόματων σταθεροποιητών και έχουμε τον Υφυπουργό Εργασίας της Ιταλίας ως υπεύθυνο συντονιστή για το ζήτημα αυτό. Ξέρουμε ότι από μόνοι μας δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σε θεσμικό επίπεδο και μη να καταφέρουν να συμβάλλουν. Διαφορετικά πολύ φοβάμαι ότι καταλήγουμε τελικά σε κάποιους παράλληλους μονόλογους όπου ο καθένας προσπαθεί να επιβεβαιώσει το ρόλο του και την πρωταρχικότητά του χωρίς να καταλήγουμε όμως σε κάποιο κοινό αποτέλεσμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να καταφέρουμε να ακολουθήσουμε αν θέλετε ένα συντονισμένο θεσμικό δρόμο. Αυτό ξεκινήσαμε να κάνουμε αυτό το εξάμεινο. Και το ξεκινήσαμε αυτό όπως σας είπα, εντάσσοντας τους κοινωνικούς εταίρους στη συζήτηση που κάναμε στην άτυπη, στο άτυπο Συμβούλιο του Μιλάνου. Κατά αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουμε μία ανταλλαγή απόψεων πολλών διαφορετικών μερών, εμπροκειμένου των κοινωνικών εταίρων, στα πλαίσια της χάραξης πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αλλάξουμε κατά κάποιο τρόπο την διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να καλύψουμε περισσότερους κλάδους και τομείς. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο απασχόλησε πάρα πολλούς στις παρεμβάσεις σας έχει να κάνει με την ανεργία των νέων, με την εγγύηση για τους νέους και τα σχετικά προβλήματα. Ω Ιταλική Προεδρία θεωρούμε ότι το ζήτημα τη ανεργία των νέων είναι πάρα πολύ σημαντικό και πειράζει προφανώ τι προπτικές τη Υπήρου μα, τι προπτικές τη Ευρώπη. Ουσιαστικά από τη δική μα την άποψη τουλάχιστον δεν μπορεί να δοθεί μία και μοναδική απάντηση. Δεν υπάρχει ένα και μοναδικό εργαλείο το οποίο θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε. Ανταυτού πρέπει να χρησιμοποιήσουμε πολλά διαφορετικά μέσα για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό. Αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό πρώτον όσον αφορά την κατάρτιση, την πρόθεση της γνώσης και της επαγγελματικής άσκησης. Δεύτερον, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η επίτευξη των απαραίτητων ποιοτικών επαγγελματικών γνώσεων. Και έπειτα η εγγύηση για τους νέους είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μέσο. Υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι οι οποίοι έχουν εγκαταλείψει τις σπουδέ τους, ενδεχομένω να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδέ τους, αλλά δεν έχουν βρει ακόμα μια θέση απασχόλησης. Το να ασχοληθούμε άμεσα με τους νέους αυτούς είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει μέσω ενός ε, ενεργητικού μηχανισμού. Θεωρώ ότι η εγγύηση για τους νέους αποτελεί ένα τέτοιο μηχανισμό. Δεν μπορούμε να περιμένουμε από το δημόσιο τομέα να καλύψει όλους αυτούς τους νέους. Δεν μπορούμε να περιμένουμε από το δημόσιο τομέα να θεσπίζει όλες τις πολιτικές. Αντίθετα, νομίζω ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε μέσα τα οποία να εμπλέκουν πιο ενεργά τους ίδιους τους νέους. Αυτό ακριβώς θέλουμε να κάνουμε μέσω της εγγύησης για τους νέους. Να καταφέρουμε δηλαδή να εντάξουμε πιο ενεργά τους νέους και στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας. Ως προς αυτό λοιπόν, εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να εργαστούμε συστηματικά για την εγγύηση των νέων και να καταφέρουμε να χρηματοδοτήσουμε καταλήλως αυτή την πρωτοβουλία. Τώρα, από πού θα προέλθει η χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση αποτελεί σαφώ προτεραιότητα, ακόμα και σε μια δεινή οικονομική περίοδο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να βρεθούν οι απαραίτητοι πόροι. Πέρα όμως από το ζήτημα αυτό, αναφερθήκατε επίσης ε, με απόλυτη σαφήνεια και στο ζήτημα της καταπολέμησης της φτώχειας. Σαφώς και αυτό το ζήτημα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο και ιδιαίτερα σημαντικό. Η συζήτηση που κάναμε στο άτυπο συμβούλιο του Μιλάνου μας επέτρεψε να συνειδητοποιήσουμε το εξής. Η στρατηγική Ευρώπη 2020 πρότεινε να μειώσουμε κατά 20 εκατομμύρια τον αριθμό των ατόμων, των απόρων ουσιαστικά, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την οικονομική όμως κρίση βρεθήκαμε ακριβώς στο αντίθετο αποτέλεσμα. Ο αριθμός των φτωχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλο αυξάνεται και προφανώς δεν μειώνεται. Θα μπορούσαμε λοιπόν να διεξάγουμε μια ολόκληρη συζήτηση για να δούμε τελικά αν οι δείκτες που αποφασίσαμε πριν από 10 χρόνια στην ε, στη Στρατηγική Ευρώπη 2020 είναι όντως οι σωστοί δείκτες. Από την άλλη μην ξεχνάμε ότι και η ίδια οικονομική κρίση επηρέασε τα πράγματα. Είναι σημαντικό πάντως να καταφέρουμε να έχουμε τις κατάλληλες κοινοτικές πολιτικές απόλυτα ευθυγραμμισμένες και συντονισμένες με τις εθνικές πολιτικές. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να δημιουργήσουμε τελικά πολιτικές ενεργούς συμμετοχής. Δεν μπορούμε να επιλύσουμε το πρόβλημα αυτό μόνο μέσω της μεταφοράς χρημάτων και κονδυλίων. Και αυτό μπορεί να συμβάλλει. Προφανώς όταν δεν υπάρχουν ε, χρήματα πρέπει ορισμένες περιφέρειες να μπορούν ε, να βασίζονται στη χρηματοδότηση που τους παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό όμως από μόνο του δεν αποτελεί λύση στο πρόβλημα σε καμία περίπτωση. Δεν θέλουμε να καταλήξουμε σε μια τέτοια κατάσταση εξάρτησης τελικά που τελικά δεν θα δώσει απτά αποτελέσματα. Ανταυτού θέλουμε πολιτικές οι οποίες θα προβλέπουν κάποια μεταφορά κονδυλίων σε ένα πρώτο βραχυπρόθεσμο στάδιο, αλλά θέλουμε μακροπρόθεσμα οι πολιτικές αυτές πραγματικά να βοηθούν τους νέους και τους άπορους για να ξεφύγουν από την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Και αναφερόμαστε βέβαια επίσης στις προτεραιότητές μας και στις οικογένειες που έχουν πάρα πολλά παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να αναφερθούμε και σε αυτή την ομάδα πολιτών. Στα παιδιά δηλαδή εκείνα τα οποία πλήττονται εξαιτίας της ε, ένδυας της οικογένειάς τους. Θα μπορούσαμε όμως να αναφερθούμε και σε ένα άλλο ζήτημα το οποίο έθιξα στην παρέμβασή μου, το ζήτημα της κοινωνικής οικονομίας, της ε, υπεύθυνη συμμετοχής των πολιτών στις διάφορες πολιτικές και δράσεις. Χρειαζόμαστε ένα νέο σύστημα πρόνοιας, χρειαζόμαστε μια νέα έννοια και προσέγγιση, αν θέλετε, της ίδιας της έννοιας της κοινότητας, της αλληλεγγύης. Και θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η σχέση μεταξύ κράτους και αγοράς δεν θα είναι η μόνη σχέση η οποία θα αποτελεί σημείο αναφοράς, αλλά θα πρέπει να υπόκειται σε συγκεκριμένες κοινωνικές συνθήκες η σχέση αυτή. Η σχέση κράτους και οικονομικής αγοράς θα πρέπει να υπόκειται σε συγκεκριμένες κοινωνικές προϋποθέσεις. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορεί ο κάθε πολίτης αλλά και κάθε επιχείρηση αν θέλετε κοινωνικά και υπεύθυνα να συμμετέχει στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση. Και ένα άλλο σημαντικό γεγονός, η, α, ο πλουραλισμός αν θέλετε των διαφόρων μορφών πολιτικών που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να επιβάλλουμε εμείς κατά προτεραιότητα κάποιες α, πολιτικές ή ότι θα πρέπει να προωθήσουμε συγκεκριμένου οργανισμούς συγκεκριμένους συλλόγους κτλ. Υπάρχει μια τεράστια πλειονότητα, ποικιλία αν θέλετε, οργανισμών, ενώσεων, συλλόγων που μπορεί πραγματικά να επηρεάσει και την ίδια την οικονομία αγοράς. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να καταλήξουμε σε μια οικονομία που θα είναι πραγματικά κοινωνική, σε μια οικονομία η οποία θα διέπεται από όλες αυτές τις κοινωνικές μορφές παρέμβασης. Μια τέτοια οικονομία νομίζω ότι θα αποκρίνεται καλύτερα και στις ανάγκες, τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών και προφανώς στα πλαίσια μια τέτοιας οικονομία, το κράτος πρόνοια, το σύστημα κοινωνικής προστασίας θα κατέχει πρωταρχική θέση. Θέλουμε λοιπόν την, όσο δυνατόν μια μεγαλύτερη υπεύθυνη κοινωνική συμμετοχή των πολιτών. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο θέσατε με τις παρεμβάσεις σας έχει να κάνει με την κινητικότητα. Αναφερθήκατε στους νέους εκείνους που αναγκάζουν να μετακινηθούν, να πάνε σε άλλες περιφέρειες, σε άλλες χώρες να βρουν θέσεις απασχόληση, το ζήτημα των αντικσοτήτων που πρέπει να αντιμετωπίσουν στις ξένες χώρες. Αναφερόμενοι στους Ευρωπαίους πολίτες θα έλεγα ότι ένας από τους πυλώνες Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ελευθερία κινήσεως κινητικότητα των εργαζομένων, των νέων μας προκειμένου. Δεν μπορούμε λοιπόν να θέσουμε να αμφιβόλο καθόλου το σημαντικότατο αυτό πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πυλώνα και πρέπει γι' αυτό το λόγο να διατηρηθεί. Δεν λέω ότι δεν θα πρέπει να συζητήσουμε, αν θέλετε, το βασικό αυτό πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε φορά που ένα σημαντικός πυλώνας ε, παρουσιάζει κάποιες προβληματικές πτυχές, προφανώς εμείς θα πρέπει να διεξάγουμε και μια σχετική συζήτηση. Σαφώς λοιπόν το ζήτημα της κινητικότητας πρέπει να μας απασχολήσει. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε τη συζήτηση λέγοντας ότι η κινητικότητα αποτελεί για μας θεμελιώδη αξία, αλλά ότι θα πρέπει να αποτελεί ελεύθερη συνειδητή επιλογή του ίδιου του πολίτη, να επιλέγει και όχι να αναγκάζει το πολίτης να μετακινηθεί. Με αυτό συμφωνώ. Όταν εξαναγκάζεται ουσιαστικά ο πολίτης να μετακινηθεί προς άλλη χώρα εξαιτίας αντιξωτήτων που αντιμετωπίζει στη χώρα του σε σχέση με κάποιες άλλες χώρες, όταν αναγκάζεται να κάνει κάτι τέτοιο λόγω της έντονης μισθολογικής διαφοράς, τότε καταλαβαίνουμε βέβαια ότι αυτό δεν αποτελεί συνειδητή ελεύθερη επιλογή του πολίτη, αλλά τελικά αποτελεί μια μορφή εξαναγκασμού, καταναγκασμού. Οι Ευρωπαίοι λοιπόν πολίτες θα πρέπει να χαίρουν ενό συστήματος ε, προστασίας οπουδήποτε και αν βρίσκονται, οπουδήποτε και αν εργάζονται. Και θα πρέπει στα πλαίσια του συστήματος αυτού να λάβουν υπόψη τα προβλήματα αλλά και τις ευκαιρίες που παρέχουν τόσο οι χώρε καταγωγή και προέλευση αυτών των εργαζομένων, όσο και οι χώρε προορισμού αυτών των εργαζομένων. Γιατί ξέρετε, τα τελευταία χρόνια αυτό που έχουμε δει είναι ότι φύστανται προβλήματα και ευκαιρίε παράλληλα και για τι χώρε προέλευση αλλά και για τι χώρε προορισμού. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι το ζήτημα αυτό είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο και λεπτό, ιδίω σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης, αλλά ουσιαστικά έχει ένα πολύ σημαντικό σημείο αναφοράς, στο ότι θέλουμε να εξασφαλίσουμε και να διατηρήσουμε τη βασική αυτή αρχή της κινητικότητας, την ελευθερία της κινητικότητας. Και κάποιος, αν δεν κάνω λάθος, αναφέρθηκε και στο ζήτημα της μετανάστευσης. Σίγουρα η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταφέρει να έχει τη δική της κοινοτική πολιτική μετανάστευση. Γιατί αυτοί οι οποίοι λένε ότι οι μετανάστες θέτουν εν κινδύνο τις θέσεις απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, θα πρέπει να ξέρετε ότι συγκυριακά δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Μπορεί να ισχύει ενδεχομένω σε κάποιες χώρες μονομένα. Αν δούμε όμως τα δεδομένα που έχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συνειδητοποιούμε ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν πάρα πολλούς μετανάστες, αλλά και υψηλότατο επίπεδο απασχόλησης. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η κατάσταση που να ισχύει συγκυριακά σε κάποιες χώρες σε καμία περίπτωση δεν φωτογραφίζει τη γενική κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν κατά περίπτωση να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν με τη μετανάστευση χωρίς να καταλήγουμε στη συνέχεια εύκολα σε γενικόλογε αποφάσει. Επίσης νομίζω ότι έχουμε μια κάποια ηθική, ιδεοντολογική υποχρέωση να αποδεχθούμε τους μετανάστες αυτούς. Σε καθημερινή βάση βλέπουμε να διεξάγονται πραγματικά δράματα, τραγωδίες με τα μεταναστευτικά ρεύματα. Έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι νετούνται σε άσυλο. Δεν μπορούμε να διαφορήσουμε απέναντι στους ανθρώπους αυτούς. Είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε κατά αυτόν τον τρόπο να τους αποκλείσουμε. Αν τους αποκλείσουμε τότε πραγματικά θα διαπράξουμε ένα πολύ μεγάλο σφάλμα και σε καμία περίπτωση δεν θα επιλύσουμε το πρόβλημα της μετανάστευσης. Συμφωνώ λοιπόν ότι ε, δεν θα πρέπει να δημιουργήσουμε νέα σύνορα και εμπόδια στα κράτη-μέλη όσον αφορά τους μετανάστες. Όταν προκύπτουν προβλήματα, αυτά θα πρέπει κατά περίπτωση να τα αντιμετωπίζουμε. Ένα άλλο ζήτημα στο οποίο νομίζω ότι αναφέρθηκαν πολλοί ευρωβουλευτέ και δεν μπορώ να καλύψω όλα τα ζητήματα που σας είπα, είναι το ακόλουθο. Έχει να κάνει με τον ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θα ήθελα να πω κάτι πάρα πολύ ουσιαστικό σε σχέση με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις αυτές διαδραματίζουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο όσον αφορά την πολιτική απασχόληση. Αποτελούν πραγματικά τη ραχοκοκαλιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος μας όμως θα πρέπει να είναι να μειώσουμε τα εμπόδια, να καταρρύψουμε τα εμπόδια τα οποία υφίστανται αυτή τη στιγμή και όχι τόσο πολύ να ασχοληθούμε με τα κίνητρα. Σαφώς εμείς θα πρέπει να βοηθήσουμε αυτές τις επιχειρήσεις. Αλλά πολύ συχνά αυτό το οποίο κάνουμε είναι ότι έχουμε μια πολιτική αντιφατική. Κάνουμε δύο πράγματα παράλληλα τα οποία είναι αντιφατικά. Βοηθούμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δίνουμε κίνητρα και χρηματοδότηση και από την άλλη δημιουργούμε περισσότερα εμπόδια και ένα μεγαλύτερο γραφειοκρατικό άχθος. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε αυτόν τον αντιφατικό τρόπο. Πρέπει σε μια πρώτη φάση να καταρρύψουμε όλα τα εμπόδια τα οποία εφίστανται αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ας μην δημιουργούμε περισσότερες δυσκολίες για τις επιχειρήσεις αυτές. Αναφερθήκατε σε αυτή την υπερβολική ρύθμιση, στη δημιουργία όλο και περισσότερων επαχθών ρυθμιστικών πλαισίων. Ας καταρρύψουμε πρώτα τα προβλήματα αυτά και νομίζω ότι αν το πετύχουμε αυτό θα έχουμε ήδη βοηθήσει πάρα πολύ τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Διατρέχω γρήγορα τις σημειώσεις μου για να δω αν απάντησα στις περισσότερες τουλάχιστον ερωτήσεις. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα το οποίο τέθη είναι η ανάπτυξη της αγοράς εργασίας στην Ευρώπη και το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το δίκτυο EURES, τις υπηρεσίες απασχόλησης δηλαδή. Και αυτό το ζήτημα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξεκινάμε ήδη αυτή τη στιγμή από μια πρωτοβουλία η οποία έχει μια πολύ σημαντική εμπειρία από πίσω της, μια πολύ επιτυχημένη ήδη ιστορία. Αυτή τη, ξεκινάμε αυτή τη στιγμή μια νέα φάση στην οποία λέμε ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε αυτές τις υπηρεσίες απασχόλησης τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για να το πετύχουμε όμω αυτό, θα πρέπει να διασυνδέσουμε το δίκτυο ΕΟΡΕΣ με ένα άλλο ζήτημα, το οποίο το θίξατε πάρα πολλέ φορέ, με το ζήτημα των γνώσεων, των δεξιοτήτων και τη αντιστοίχηση ανάμεσα στι δεξιότητε και τι πραγματικέ ανάγκε και προσφορέ αγορά-εργασία. Θα πρέπει εμεί να χρησιμοποιήσουμε τα κατάλληλα εθνικά και ευρωπαϊκά μέσα τα οποία θα πρέπει να είναι συντονισμένα και τα οποία θα μας επιτρέψουν να έχουμε μια ευθυγραμμισμένη στρατηγική ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κατάλληλες, κατάλληλες τράπεζες δεδομένων, για παράδειγμα τα κατάλληλα προγράμματα κατάρτισης για την επίτευξη των πιο ευκταίων δεξιοτήτων. Να καταφέρουμε δηλαδή να δώσουμε ιδίω στου νέου που μετακινούνται πιο εύκολα τι απαραίτητε πληροφορίε, την κατάλληλη ενημέρωση. Η εργασία λοιπόν που θέλουμε να επιτελέσουμε στα πλαίσια του ΕΟΡΕΣ είναι ακριβώς αυτή, να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο δεύτερης γενιάς, λαμβάνοντας υπόψη μας το ότι υπάρχουν πάρα πολλές χώρες οι οποίες μας είπαν και μας λένε συνεχώς ότι έχουν ένα υψηλότατο επίπεδο γραφειοκρατίας. Μέσω λοιπόν του δικτύου ΕΟΡΕΣ μπορούμε να αποφύγουμε ή θα πρέπει τουλάχιστον να αποφύγουμε να δημιουργήσουμε ένα νέο επίπεδο υπερβολικής ε, ρύθμισης. Ας εργαστούμε λοιπόν στα πλαίσια του ΕΟΡΕΣ προκειμένου να έχουμε μια ευθυγραμμισμένη στρατηγική για την αγορά εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς όμως να καταλήξουμε σε επικαλύψεις, χωρίς ε, να δημιουργούμε περιττές νέες ρυθμίσεις. Είμαι βέβαιος ότι δεν απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις σας, αλλά ενδεχομένω θα ήταν αδύνατο να κάνω και κάτι τέτοιο, δεδομένου του χρόνου. Ολοκληρώνω πάντως ε, ευχαριστώντας για άλλη μια φορά την Επιτροπή σας ε, για όλες αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις και παρατηρήσεις. Έχω καταγράψει όλα τα μελήματά σας, όλες τις ερωτήσεις σας, όλες τις παρατηρήσεις σας και είναι καθήκον μου να χρησιμοποιήσω τις παρατηρήσεις αυτές στις εργασίες τις οποίες θα επιτελέσω στα πλαίσια του Συμβουλίου. Όπως σας είπα είμαι στην πλήρη διάθεσή σας προκειμένου να έχουμε μια επικοδομητική συνεργασία γιατί θεωρούμε ότι η συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τη δική μας την Προεδρία είναι αν θέλετε ο καλύτερος δυνατός τρόπος για να αντιμετωπίσουμε τα σημαντικότητα αυτά προβλήματα που έχουμε στο τομέα της απασχόλησης. Μέσω της επικοδομητικής αυτής συνεργασίας θα καταφέρουμε να βρούμε κοινέ λύσεις, λύσεις οι οποίες θα προκύψουν μέσω του κοινού διαλόγου. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ελπίζω ότι δεν σας απογοήτευσα, ότι ανταποκρίθηκα έστω και λίγο στι προσδοκίε σα. Λυπάμαι, οι ερωτήσει ήταν πάρα πολλέ, ιδιαίτερα ευρύς και ενδεχομένω να μην κατάφερα να απαντήσω σε όλες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργή. Σίγουρα σε 22 ερωτήσεις δεν μπορείτε να απαντήσετε. Το κατανοώ αυτό, αλλά πρωτού φύγετε να, να δείξω τρία σημεία. Έδειξε η συζήτησή μας ότι αυτή η Επιτροπή είναι δεσμευμένη να εργαστεί σε θέματα απασχόλησης στη συνεδρίαση των συντονιστών είπαμε ότι θα πρέπει να συμμετέχουν και άλλοι φορεί στη συζήτηση αυτή. Επίσης, ε, η ενδιάμεση αξιολόγηση για τη Στρατηγική Ευρώπη 2020, ε, η οποία θα είναι έτοιμη και αυτά πρέπει να συζητηθεί. Ξεκινάμε από σήμερα λοιπόν τις εργασίες μας και όλα αυτά βέβαια θα τα δούμε σε συνάφεια με την Ιταλική Προεδρία. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε για το TTIP. Θα μας απασχολήσει το θέμα αυτό και θα γίνει μια ακρόαση το φθινόπορο σε σχέση με τα εργασιακά δικαιώματα στο πλαίσιο πάντα του, της Ιταλικής Σχέσης Συναλλαγών και Επενδύσεων. Μια παράκληση σας κύριε Υπουργέ. Οι θυμίσεις που έχουν γίνει από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, προστασία των μητέρων να μην ε, εκμεταλλεύονται, να γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευση και να μην επιβαρύνονται με υπερβολική ε, γραφειοκρατία. Σε ένα διάλειμμα μετά τη συνεδρίαση αυτή θα μπορούσα να το παρουσιάσω αυτό καλύτερα, ειδικά όσον αφορά ε, τον έλεγχο των αποσπασμένων εργαζομένων. Η βούληση του εργοδότη είναι πολύ σημαντική, ειδικά ε, έχοντας υπόψη ένα πρόγραμμα ε, αποφυγής κατάρχησης της γραφειοκρατίας όπως είναι το REFIT. Σας παρακαλώ λοιπόν όλους να δεσμευτείτε ώστε να γίνει κατανοητό ότι δεν αποφασίζουμε για κλεισμένο του θυρών. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για την επισκεψή σας. Θα είμαστε σε επαφή ε, για να συζητήσουμε και για αυτά τα, τα φλέγοντα κοινωνικά θέματα και θα ε, υποστηρίξουμε την Προεδρία. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. So, Kolleginnen und Kollegen, darf ich bitte... Συνάδελφοι, συναδέλφες, καθίστε και πάλι. Wir werden dann bei Tagesordnungspunkt 4 des Budget der Europäischen Union für das Θα περάσουμε στο σημείο 5 ε, Προεπιλογής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015. Ε, Ανταλλαγή απόψεων είχαμε σε πρώτη ε, φάση το πρόβλημα είναι ότι το έγγραφο εξαιτία του λίγου χρόνου που έχουμε στη διάθεσή μας δεν είναι μεταφρασμένο σε όλες τις γλώσσες, το έχουμε μόνο στα αγγλικά. Αλλά θεωρώ ότι για μια πρώτη ανταλλαγή ε, απόψεων μπορούμε να βαστούμε σε αυτό το αγγλικό κείμενο. Μας λείπει αρμοδιότητα, δεν έχουμε την αρμοδιότητα στην Επιτροπή για αυτό το θέμα. Θα προετοιμάσουμε αυτή τη γνωμοδότηση, η οποία θα αποσταλεί στη συνέχεια στην Επιτροπή Υπροπολογισμού. Η Μαρία Αρένα από το S&D είναι η συγγήτρια. Μπορεί να μας παρουσιάσει αυτή την πρόταση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να πω ότι η πρόταση αυτή είναι πολύ καλή. Η Μαρία Αρένα θέτει προτεραιότητες ώστε οι απλήρωτοι λογαριασμοί ε, να, πλη, να, κατα, να πληρωθούν. και ότι θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη και το 2015 το θέμα της ενεργείας στο νέα. Προτάθηκαν πολύ λίγα χρήματα από την πλευρά του Συμβουλίου. Αυτό το, συζητήσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Προτάθηκαν όμως και άλλες αναγκαινότητες οι οποίες θα πρέπει να ενταχθούν στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Η κυρία Αρένα, η συγγήτρια, προτείνει πιλωτικά προγράμματα, μια ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης, Και αυτά είναι αποτέλεσμα ε, μια έκθεσης που κάναμε μαζί πέρσι. Και προτείνει λοιπόν ένα επιλογικό πρόγραμμα για την ενέργεια, για τη φτώχεια, ε, μέτρα για τον αμίαντο, Όλες πολύ καλές οι προτάσεις. Η συγκήτρια περιμένει και τα σχόλια των συναδέλφων στην Επιτροπή. Και φυσικά αν έχετε ερωτήσεις μπορώ να τις απαντήσω. Ευχαριστώ Γιώτα ε, Στάιντρουκ. Ο σκιώδης συγγητής ε, Μάρκ Μυρόσλαβ Πλούρ από το ΕΛΚ θα μιλήσει στη συνέχεια. Ως σκιώδης συγγητής θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Μαρία Αρένα για την παρουσίαση αυτής της γνωμοδότησης για το σχέδιο Πολιτισμού του 2015. Συμφωνώ πλήρως με την προσέγγιση της ότι θα πρέπει αυτός ο προπολογισμός να δημιουργηθεί βασικό ρόλο στην ανάπτυξη και στην απασχόληση και στην βελτίωση συγκεκριμένα της δυσχερούς ε, κατάστασης των ε, νέων στην αγορά εργασίας. Είναι απαραίτητο λοιπόν να διασφαλίσουμε πλήρη πρόσβαση σε οικονομικά μέσα υπό την πρωτοβουλία για τις εγγύσεις των νέων και, ε, για το Ευρωπαϊκό, και υπό το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Έχουμε βιώσιμες αλλαγές στην αγορά εργασία. Θα θέσουμε τις σωστές συνθήκες για τη δημιουργία μικρομεσαίων επιχειρήσεων που προσφέρουν το 65% των ε, θέσεων απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι λοιπόν στις τροπολογίες μου θα θέλω να δώσω έμφαση ότι πρέπει να χρηματοδοτήσουμε επαρκώς τις ε, νεοφυείς επιχειρήσεις για να υποστηρίξουμε την δημιουργία μικρομεσαίων επιχειρήσεων και φυσικά να μειώσουμε και την γραφειοκρατία. Είναι πολύ σημαντικό να προωθήσουμε, να προάγουμε την ε, κοινωνική επιχειρηματικότητα και τα ε, μικροδάνεια. Για να ξεπίσουμε το δυναμικό μας σωστά πρέπει να δώσουμε ισότιμες ευκαιρίες ε, στους, ε, στα άτομα με ειδικές ανάγκες και να διασφαλίσουμε πρόσβαση στην αγορά εργασίας και σε αυτούς. Υπάρχει ψηλό ποσοστό φτώχειας, φτώχεια ε, στην παιδική ηλικία και γι' αυτό πρέπει να παρέχουμε τα οικονομικά μέσα για αυτούς που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Η γνωμοδότηση της Επιτροπής μας θα πρέπει να αντικατοπτρίζει αυτές τις προτεραιότητες που έχουμε σε σχέση με αυτά ε, μιλάω συγκεκριμένα για τον προπολογισμό του 2015. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσει ο κύριος Τρεμπέζιος εκ μέρους του ECR. Κυρία Τρεμπέζιος. Έχει φύγει από την αίθουσα, λοιπόν. Μαρίαν Άρκιν, εκ μέρους του Άλντε. Ευχαριστώ και ευχαριστώ την εισηγήτρια για την καλή της δουλειά σε αυτή την γνωμοδότηση. Υποστήριξα τις προτάσεις της. Όσον αφορά την τοποθέτηση του Συμβουλίου για τον προπολογισμό, λάβαμε την εξή πληροφόρηση σήμερα και δεν είχα χρόνο να την ερευνήσω. Θα το κοιτάξω πιο καλά αργότερα, όσον αφορά τις προτάσεις της συγκήτριας, τις υποστηρίζω πλήρως. Και συγκεκριμένα εκεί που κάνει αναφορά για την εγγύηση των νέων, θα μπορούσε αυτό να διατυπωθεί με πιο επιτακτικό τρόπο ενδεχομένω. Επίσης, ε, σε σχέση με το EGF, είχαμε αιτήσει και γι' αυτό το οποίο είναι ενθαρρυντικό γιατί δεν είναι το ταμείο το οποίο μπορεί να βοηθήσει στον τομέα της ενεργείας των νέων πλέον. Θα ήθελα να ενθαρρύνω τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα όταν τους δίνεται και όσον αφορά τα πιλωτικά προγράμματα, τα υποστηρίζω και αυτά. Δεν έχω πολλά άλλα να προσθέσω, απλώς να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την ε, δουλειά της. Ευχαριστώ από τον Γκουε τώρα. Όχι, μάλλον περνάμε στους πράσινους. Ντάμας Μέσεριτς. Ευχαριστώ πολύ. Ε, εγώ είμαι αναπληρωτής, δεν είμαι πλήρες μέλος. Ευχαριστώ τους εισηγητές, υποστηρίζουμε τις βασικές ιδέες οι οποίες ε, υποβλήθηκαν και νομίζω ότι έχουμε λογικό συμβιβασμό για ορισμένα θέματα που αναφέραμε Συμφωνώ επίσης πλήρως ότι ε, η εμπροστοβαρής προσπάθεια είναι καλή ιδέα. Υπάρχει ε, καμιά, είναι καλή ιδέα, αλλά όχι να μην ε, χρησιμοποιείται υπερβολικά. Καμιά φορά δεν έχει καλά αποτελέσματα. Πρέπει να δούμε πώς απορροφώνται τα, τα, τα, τα, τα κονδύλια αυτά για μεγάλα έργα, διότι πάρα πολλοί δεν έχουν την ικανότητα απορρόφησης πολλά κράτη-μέλη δέχομαι που δεχτήκατε την πρόταση για το πιλωτικό πρόγραμμα για την ε, φτώχεια. Ελπίζω ότι θα είναι από τα βασικά θέματα της ε, τα επόμενα χρόνια. Είναι κάτι περισσότερο από αυτό που φαίνεται εκ πρώτης όψεως και ίσως να είναι ένα θέμα σημαντικό αργότερα. Βλέπουμε επίσης ότι υπάρχουν μικρές συμβολικές περικοπές σε ορισμένες γραμμές του προϋπολογισμού ε, που θα θέλαμε ε, να μην γίνουν για να κρατήσουμε το συμβολισμό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. το αυτή δεν έχουμε ε, εισηγητή. Μήπως υπάρχει κάποιος που θα θέλει να μιλήσει εκ μέρους του ΕΦΔ. Όχι, οπότε... Συνεχίζουμε. Δεν μπορώ να διαβάσουμε στο το όνομα του επόμενου μιλητή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι η πρόταση να έχουμε ε, μια κάρτα ασφαλείας ε, ευρωπαϊκή ε, είναι ένα σύστημα ταυτότητας ευρωπαϊκής ενιαίας δεν είναι. Ε, και έτσι οι εθνικές κυβερνήσεις δημοκρατικά εκλεγμένες ε, θα, ε, θα αντιδεθούν σε πιο συγκεντρωμένη εξουσία στις Βρυξέλλες. Θα έχουμε, είχαμε με την ιδέα αυτή μεγάλη οργή που εκφράστηκε στην, στο Ηνωμένο Βασίλειο και πώς οι πολλές πληροφορίες για την κάρτα θα αποθηκευθούν. Τέθηκαν πάρα πολλά ερωτήματα και πώς θα χρησιμοποιούνται. Οποιαδήποτε πληροφορία που σχετίζεται με την Ευρωπαϊκή Κάρτα θα πρέπει να ενημερώνεται και όταν το σύστημα καθιερωθεί πόσο περισσότερες πληροφορίες θα απαιτούνται στο μέλλον. Κάθε πρόβλημα αυτού του είδους έχει επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα, κυρίως όταν η ανάγκη ασφάλειας θα απαιτεί οι πολίτες να παρέχουν βιομετρικά δεδομένα και στοιχεία. Και το κόστος ενός τέτοιου προγράμματος πριν πέντε ε, χρόνια όταν ακυρώθηκε το πρόγραμμα της Βρετανίας, αξιολογήθηκε σε περίοδο 10 ετών ότι θα κόστιζε 800 εκατομμύρια για να καλυφθούν 65 εκατομμύρια άτομα. Όταν ε, προβάλλουμε τον αριθμό ε, σε 500 ε, εκατομμύρια θα έχουμε 6 δισεκατομμύρια. Όποια αύξηση πληθωριστική θα είναι επίσης απειλή απειλή για την ασφάλεια. Ωστόσο, είναι η συλλογή των φορολογικών στοιχείων ε, των πολιτών που είναι ανησυχητική. Θα είναι δύσκολο να γίνει αυτό ε, χωρίς ε, να υπάρχει μια πολιτική ενιαία συγκεντρωτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, θα είναι περαιτέρω βήματα για την εκπλήρωση του ονείρου του κυρίου Γιούνκερ για ένα υπερκράτος ευρωπαϊκό. Και αυτό νομίζω συγκαλύπτει τις πραγματικές προθέσεις του από τους ψηφοφόρους. Ευχαριστώ. Έχουμε ακόμα έναν ομιλητή, την κυρία Νατώνα Σανοβιέτσκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η γνωμοδότηση αφορά χρήματα. Ε, όταν κάνουμε λόγο για την ενεργεία των νέων και την καταπολέμησή της, με ικανοποιεί, με ικανοποιεί αυτή η στήριξη πιλωτικών προγραμμάτων, δεδομένης και της δύσκολης κατάστασης με τους μετανάστες. Στην Ευρώπη επίσης θα ήθελα να προτείνω μια τροπολογία καθώς θα υποστηρίξουμε την ιδέα κέντρων υποδοχής, υποστήριξης για τους μετανάστες, ώστε να τους παρασχεθεί βοήθεια για να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Ο λόγος ε, στην Επιτροπή στον Όλιβερ Ρουλάντ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι αρκετά σύντομος. Πρώτα απ' όλα ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτήν τη γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου που τίνει να αποκαταστήσει την πρόταση της Επιτροπής κατά κάποιο τρόπο ακόμη και πάνω σε ένα σημαντικό σημείο το οποίο δεν περιλαμβάνεται στο σχέδιο γνωμοδότησης. Είναι η πρώτη φορά που προτείνεται μια περικοπή των πιστώσεων υποχρεώσεων και επισύρω την προσοχή σας πάνω στο θέμα αυτό, ενώ ψηφίστηκαν οι δημοσιονομικές πρόπτικες. Επισύρω την προσοχή σας πάνω στο θέμα αυτό σχετικά με τα πιλωτικά έργα πρώτου κύματος υπήρξε μια αντίδραση επίσημη της Επιτροπής που τίνει στο να επισύρει την προσοχή πάνω στο γεγονός ότι τα θέματα είναι σημαντικά και ε, Επίση να επισύρει την προσοχή του Κοινοβουλίου πάνω στην ε, συμπερίληψη την ε, σημαντική του θέματος αυτό στα προγράμματα τα υφιστάμενα εργασίας. Είναι ένα σημείο το οποίο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στην πρόταση πιλωτικών προγραμμάτων. Και είναι αυτή η άποψη σημαντικότερη που χρησιμοποιούμε. Είναι ήδη, καλύπτεται ήδη ή όχι από τις νομικές υφιστάμενες βάσεις, ε, τους υφιστάμενους προϋπολογισμούς. Ε, αυτά. Αυτό είναι το ερώτημα. είναι σκόπιμο ή ενδιαφέρον ε, να αφιερώσουμε περισσότερους πόρους σε αυτόν τον προβληματισμό. Δεν ξέρω για τα θέματα, τα ιδιαίτερα, ιδιαίτερα θέματα, αν θέλετε, να διευκρινίσω κάτι ως Επιτροπή. Υπάρχουν ερωτήσεις ε, στην Επιτροπή. Αν όχι, θα δώσω και πάλι το λόγο στην ε, αντικαστάτρια της ε, εισηγήτριας. Η συνάδελφός μου, η Μαρία Ρένα, θα χαρεί πολύ για την υποστήριξη που έχει η γνωμοδότησή της. Με παρακάλεσε να σας εξηγήσω ότι θα προσθεθεί ακόμα ένα πιλωτικό πρόγραμμα για το ελάχιστο εισόδημα. Τα πολιτικά προγράμματα δεν είναι εφαρμογή, αλλά η δοκιμή ενδεχόμενων μέτρων όσον αφορά την χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτό δεν μας αφορά εδώ στην Επιτροπή. Αυτό είναι θέμα της ε, Ήτρα. Επομένως είναι λίγο δύσκολο να το συμπεριλάβουμε στην γνωμοδότησή μας θα χαρεί όπως και να έχει να συνεργαστεί με τους κοιόδης συγητές και ε, να μελετήσει τις ε, προτάσεις για τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ. Äh, λοιπόν, συνεχίζουμε. Η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι 25 Ιουλίου, 12 η ώρα το μεσημέρι. Αποκλειστικά σε αγγλικά οι προτάσεις. Επειδή έχουμε μόνο την εγγλική εκδοχή του κειμένου, παρακαλούμε και οι τροπολογίες να είναι στα αγγλικά. 25 Ιουλίου, λοιπόν, του 2014, στις 12 το μεσημέρι. 3 Σεπτεμβρίου θα μιλήσουμε για τις ε, τροπολογίες και θα ψηφίσουμε για αυτή την ε, έκθεση. Στι 4 Σεπτεμβρίου είναι η ψηφοφορία στην Επιτροπή Προπολογισμού. Μάλλον 1η Οκτωβρίου θα γίνει η ψηφοφορία. Η προθεσμία για τροπολογίε στην Επιτροπή Βάτσαντη είναι μέχρι 4 ε, ε, Σεπτεμβρίου. Αυτά λοιπόν και περνάμε στο σημείο τη μερική διάταξη, το σημείο 5, η δημιουργία Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για τη συνεργασία ενάντια στην αδήλωτη εργασία για την πρόληψη και την πάταξη της αδήλωτης εργασίας. Πρέπει να ορίσουμε εισηγητή. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε σήμερα, να ανταλλάξουμε απόψεις με τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στις 9 Απριλίου υιοθέτησε αυτή τη θέση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμείς ε, θα ορίσουμε εισηγητή τον Σεπτέμβριο. Αυτή είναι μία από τις βασικές πρωτοβουλίες, όπως είναι γνωστό, ε, μία από τις προτεραιότητες της ε, Ιταλικής Προεδρίας. Ελέγχθηκε η πρόταση από την ΕΟΚΕ, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ήδη. Οπότε σήμερα μπορούμε να έχουμε μια αρχική συζήτηση επί του θέματος με τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κύριο Μούρι Γκουίν. Ο λόγος σε αυτόν. Merci Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, ένας Ευρωπαίος στους 10 αποδέχθηκε ότι έχει αγοράσει προϊόντα ή υπηρεσίες προκύπτουν από την αδήλωτη εργασία και ένα 4% των ερωτηθέντων παραδέχθηκε ότι ασκούσε αδήλωτη εργασία. Ξέρουμε όλοι μας ότι η αδήλωτη εργασία παίρνει διάφορες μορφές, διαφορετικές μορφές, ανάλογα με το κράτος μέλος, αλλά ουσιαστικά είναι ένα φαινόμενο το οποίο επηρεάζει όλα τα κράτη-μέλη και έχει πολύ δυσμενείς συνέπειες για τους ίδιους εργαζομένους, για τις επιχειρήσεις, αλλά και για την κοινωνία στο σύνολό της, καθώς επίσης και για τους εθνικούς ε, προϋπολογισμούς. Πρόκειται λοιπόν για μια πρόκληση που αφορά όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης. Οι αρνητικές αυτές συνέπειες εντοπίζονται προφανώς στις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων, ιδίως όσον αφορά το ζήτημα της κοινωνικής υγειονομικής κάλυψης στον χώρο εργασίας, αλλά ουσιαστικά έχει να κάνει και με κάποια δικαιώματα των εργαζομένων, όπως οι άδειες, ο χρόνος εργασίας, το δικαίωμα σε κατάρτιση, ή επηρεάζει επίσης και το ζήτημα της ασφάλισης της εργασίας, το ζήτημα των επιδομάτων ανεργίας και το καθεξής. Αρνητικές επίσης είναι και οι επιπτώσεις όσον αφορά την βιωσιμότητα των συντάξεων των ατόμων που βρίσκονται σε κατάσταση αδήλωτης εργασίας και προφανώς υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις και στον ανταγωνισμό. Αρνητική λοιπόν η επίπτωση σε εθνικό επίπεδο, ιδίως όσον αφορά τα φορολογικά έσοδα και ιδίως όσον αφορά τις κοινωνικές εισφορές. Κατά αυτόν τον τρόπο μειώνεται ο εθνικός προπολογισμός και η δυνατότητα των κρατών μελών να θεσπίσουν ενεργές πολιτικές και να χρηματοδοτήσουν τέτοιες πολιτικές στον τομέα της απασχόλησης. Σε κοινοτικό επίπεδο συνέβησαν τελευταία χρόνια κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Πολλά κράτη-μέλη συσπυρώθηκαν σε επιμέρους ομάδες για να δουν τι θα μπορούσαν να κάνουν προκειμένου να αντιμετωπίσουν συλλογικά το ζήτημα της αδήλωτης εργασίας. Αυτό το οποίο συνειδητοποίησαν όμως είναι ότι δεν υπάρχει κάποιο όργανο, κάποιο φόρουμ, μια οντότητα αν θέλετε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα επέτρεπε μια πραγματική επικοδομητική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών για την πάταξη της αδήλωτης εργασίας. Δεν υφίσταται λοιπόν σφαιρική ολιστική προσέγγιση, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι υπάρχουν κάποια κρατημέλη που ασχολούνται κυρίως με τις συνθήκες εργασίας, άλλα κρατημέρια που ασχολούνται με την κοινωνική ασφάλιση δεν υπάρχει μία κοινή δεξαμενή γνώσεων και εμπειριών όσον αφορά την πάταξη του φαινομένου αυτού. Και κατά αυτόν τον τρόπο τα κράτη-μέλη δεν καταφέρνουν επικοδομητικά να αντιμετωπίσουν κυρίως τις διασνοριακές πτυχές της αδήλωτης εργασίας. Βάσει λοιπόν της διάγνωσης αυτής, το ότι δηλαδή η αδήλωτη εργασία παίρνει διάφορες μορφές και ότι αποτελεί προφανώς κοινό πρόβλημα για όλα τα κράτη-μέλη, και μετά τη συνειδητοποίηση επίσης από τα κράτη-μέλη ότι το φαινόμενο αυτό υφίσταται και ενισχύεται, μολονότι έχουν καταβληθεί κάποιες προσπάθειες και αναλήφθησαν κάποιες πρωτοβουλίες από ορισμένα κράτη-μέλη τα τελευταία χρόνια. Μετά από όλα αυτά λοιπόν εμείς αποφασίσαμε στις 9 Απριλίου να δημιουργήσουμε μία πλατφόρμα με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας για την πρόληψη και την αποτροπή της αδήλωτης εργασία. Πλατφόρμα λοιπόν συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών που επιτρέπει τη συμμετοχή όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω των εθνικών τους αρχών και συγκεκριμένα των αρχών ελέγχου και επιτήρησης ε, της ε, εργατικής νομοθεσίας. Αυτοί που εργάζονται μέρα με την ημέρα ε, και δουλεύουν αδήλωτα σε μαύρη εργασία, αποφεύγουν τις επιθεωρήσεις εργασίας, τον έλεγχο της κοινωνικής ασφάλισης κλπ να είναι ένα φόρουμ ανταλλαγής ε, τακτικό, διαρθρωτικό συνεργασίας, να αναπτυχθεί αυτή η ολιστική προσέγγιση που είναι απαραίτητη, διότι είναι ένα σύνθετο περίπλοκο πρόβλημα η αδήλωτη εργασία και θα ε, υποστηρίξουμε και θα συμπληρώσουμε ε, τις προσπάθειες των κρατών μελών στον τομέα αυτό στις εθνικές αρχές των κρατών μελών και ε, στην Κομισιό έρχεται να προσθεθεί ως παρατηρητής ε, Αυτή της πλατφόρμας, η κοινωνική εταίρη, στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπενθυμίζω ότι για να προετοιμάσουμε αυτήν την πρόταση που κατατέθηκε βάσει του άρθρου 153 η Κομισιό συμβουλεύτηκε σε δύο φάσεις τους κοινωνικούς εταίρους πράγμα που μας επέτρεψε να εμπλουτίσουμε την πρόταση με ιδέες που προέρχονται από τους κοινωνικούς εταίρους. Επίσης θέλουμε να προσθέσουμε τα ιδρύματα, το Ίδρυμα του Δουβλίνου και την ΟΤΣΑΤ, ε, του Μπιλμπάο και όπως και την Διεθνή Οργάνωση Εργασίας και μερικές χώρες ε, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Η βασική στόχη αυτής της πλατφόρμας θα είναι η καλύτερη ε, υλοποίηση των εθνικών κανόνων σε σχέση με την αδήλωτη εργασία, αλλά και των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, η δημιουργία ε, τυπικών επίσημων θέσεων εργασίας και η ένταξη στην αγορά εργασίας και η κοινωνική ενσωμάτωση και αυτό διαμέσου τριών μεγάλων στόχων που είναι η βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων εθνικών αρχών, η βελτίωση της, της, των δυνατοτήτων τους των τεχνικών ε, να ε, κατανοούν, να καταγράφουν ε, τις, τα διασυνοριακά φαινόμενα και καταστάσεις, η αύξηση ε, τους εντύπωση ότι το θέμα είναι κατεπήγον, το κοινό να αισθανθεί ότι το θέμα είναι κατεπήγον. Θα υπάρξουν τρεις αποστολές, η ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών και πληροφοριών, η ανάπτυξη πραγματογνωμοσύνης και ικανότητας ανάλυσης και ο συντανισμός ε, δράσεων επιχειρησιακών διασυνοριακών. Και προτείνουμε στον συνομοθέτη έναν αριθμό πρωτοβουλειών, εργασιών για να ε, εκπληρωθούν οι διάφοροι αυτοί στόχοι. Ε, είναι πολυπληθής στο ύψος των προκλήσεων, βεβαίως η βελτίωση της γνώσης του φαινομένου της αδήλωτης εργασίας. Όπως είπα, υπάρχουν διαφορετικές χαρακτηριστικές ανάλογα με τις εθνικές αγορές εργασίας. Υπάρχουν κρατημέλη που δεν έχουν ακόμη ε, στους ε, διάφορους ε, κώδικες τους την αδήλωτη εργασία ως αδίκημα, ειδικό αδίκημα. Θα πρέπει να βελτιωθεί αυτή η γνώση λοιπόν θα πρέπει να αναλυθεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν ληφθεί στην επίπεδο των κρατών μελών μέχρι τώρα. Θα πρέπει να αναπτυχθούν εργαλεία πρακτικά για τους επιθεωρητές εργασίας και για άλλους συναδέλφους από τις αρχές επιτήρησης και εποπτείας για να βελτιωθεί η αντίληψή τους του φαινομένου και να έχουν μέσα για να μπορέσουν να προσδιορίσουν πιο εύκολα το φαινόμενο της αδήλωτης εργασίας. Θα πρέπει να αναπτυχθούν οι μορφές διασυνοριακής συνεργασίας. Ένα σημαντικό στοιχείο είναι να εξεταστούν τα μέσα βελτίωσης των ανταλλαγών πληροφοριών και στοιχείων που απαιτούνται ανάμεσα στα κρατημέλη, τηρώντας πάντοτε την προστασία των προσωπικών δεδομένων, επίσης η ανάπτυξη δυνατοτήτων, ικανοτήτων κατάρτισης των, ε, των συναδέλφων των εθνικών αρχών και επίσης να οργανωθούν και να υποστηριχθούν εκστρατείες ευρωπαϊκές είτε οριζόντιες είτε τομεακές. Ιδιαίτερα που πλήττονται ιδιαίτερα από το φαινόμενο της αδήλωτης εργασίας. Αυτά γενικά είναι οι μεγάλοι στόχοι της πρότασης. Θα είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς να συνεργαστούμε με τον ή την εισηγήτρια που θα οριστεί από το Κοινοβούλιο. Πρόκειτο για ένα θέμα που το Κοινοβούλιο θεωρήσε πάντοτε ως σημαντικό ε, με παρακίνηση της κυρίας Στάμπρουκ το Δεκέμβριο το Κοινοβούλιο υιοθέτησε ένα ψήφισμα για πιο αποτελεσματικές στρατηγικές επιθεώρησης της εργασίας όπου η αδήλωτη εργασία θα πρέπει να τύχει ε, καλύτερης συνεργασίας. Από τις 9 Απριλίου οι συζητήσεις άρχισαν στο Συμβούλιο και έχουν ε, προχωρήσει καλά στα πλαίσια της ελληνικής προεδρίας και συνεχίζονται με την Ιταλική προεδρία, όπως το υπενθύμησε ο Υπουργός προηγουμένως. Ακόμη συζητούνται, αλλά υπήρξαν πρόοδοι το θέμα της συμμετοχής της υποχρεωτικής των κρατών μελών και επίσης υπάρχουν συζητήσεις για τις μορφές και τον κατάλογο των πρωτοβουλειών που προτείνονται από την Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Ζητούν αρκετοί το λόγο. Πρώτα η συνάδελφος Στάιμπρουκ. Ευχαριστούμε για την παρουσίαση πέρσι στο πλαίσιο της οδηγίας για τους αποσπασμένους εργαζόμενους ε, αποκτήσαμε μια πολύ αναλυτική εικόνα της κατάστασης. Γίνανε καλές προτάσεις για την καταπολέμηση της αδειλούδης εργασίας. Η κοινωνική εκμετάλλευση, η φοροδιαφυγή, και όλα αυτά έχουν, ε, οδηγούν σε πολύ μεγάλες απώλειες. 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ είναι οι απώλειες εξαιτία όλων αυτών των φαινομένων. Θεωρώ ότι η πρόταση της Επιτροπής είναι μια καλή αρχή όμως δεν ε, προχωράει αρκετά. Επίσης, θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και την ψευδή αυτοαπασχόληση. Έχετε ήδη την υπερογνωμοσύνη των ε, κοινωνικών εταίρων, αναφερθήκατε σε αυτήν και ότι μπορούν να συνεισφέρουν οι οποίοι όμω μέχρι στιγμή σε αυτή την πλατφόρμα έχουν μόνο ρόλο παρατηρητή. Αυτή η κοινωνική εταίρη είναι τα συνδικάτα που στο παρελθόν ήταν οι μοναδικοί που πραγματικά ε, κάλυψαν ε, την... Ε, ε από αυτή, την, ε, αυτά τα φαινόμενα τη ελληνική εργασία. Δεν θα πρέπει μόνο να λύσουμε το θέμα, αλλά να εντοπίσουμε και τις εταιρείες γραμματοθυρίδας και να δούμε και πώς ε, θα υπάρξει και συνοριακός έλεγχος. Και φυσικά το πιο σημαντικό είναι η δεσμευτική συμμετοχή σε αυτό το πρόγραμμα όλων των κρατών μελών, ώστε να είναι αποδοτικό ο έλεγχο. Και θα πρέπει κάθε κράτος μέλος να δεσμεύεται σε όλους τους τομείς, όχι να επιλέγει ανάλογα με τη βούλησή του θα πρέπει να δράσουμε από κοινού, να δεσμευτούμε και να δράσουμε και όχι απλά να μείνουμε στα λόγια. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος ε, στον κύριο Ζάσπαχ, στον κύριο Μπαχ. Να υποστηρίξω την Επιτροπή και να της χαρώ για αυτή την ανακοίνωση. θεωρώ ότι πρέπει να, το, να δώσουμε πολύ μεγάλη έμφαση στο θέμα της αδελφής εργασίας. Είναι πολύ μεγάλο, στο, μεγάλο το κόστος, αλλά και για τους ίδιους τους εργαζόμενους το κόστος είναι πολύ υψηλό επίσης. Η συμμετοχή σε αυτή την πλατφόρμα πρέπει να είναι δεσμευτική. Διαφορετικά, θα μείνουμε μόνο στα λόγια, θα έχουμε ένα απλό έγγραφο. Τα κράτη-μέλη αν δεν είναι δεσμευτικό αυτό το όργανο, αυτό το μέσο, τότε δεν θα δείξουν και την απαραίτητη προθυμία. Δεν είχα χρόνο το ε, μελετήσω λεπτομερώ ε, λόγω έλλειψη χρόνου. Το έγραφε αυτό, αλλά θέλω παρόλα αυτά να συγχαρώ την Επιτροπή. Ο λόγο στην ε, Σοφία Ριμπέρο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κομισιό για αυτήν την πρωτοβουλία. Σύμφωνο πλήρως ότι Χρειαζόμαστε μέτρα για την κοινωνική προστασία. Πρέπει να καταπολεμήσουμε την παράλληλη οικονομία. Συμφωνώ με όλα αυτά. Θα έλεγα όμως ότι αυτή η πρωτοβουλία θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ σημαντική ε, για τις ε, περιφέρειες που ζουν τη μεγαλύτερη κρίση. Έρχομαι από τις Αζόρες που είναι μια υπερπεριφερειακή ζώνη. Ε, σε σχέση με τον μόσο όρο είμαστε πολύ χαμηλά στις αζόρες και θα ήθελα ε, να θέσω τα ακόλουθα θέματα. Συμφωνώ ε, με, τον, με τη συνάδελφο η οποία είπε ότι δεν καταλαβαίνει γιατί τα συνδικάτα δεν έχουν μεγαλύτερο ρόλο σε αυτήν την πλατφόρμα και έχουν μόνο ρόλο παρατηρητή. Εγώ προέρχομαι από το συνδικαλιστικό κόσμο, έχω κάνει πολλή δουλειά στο θέμα και δεν καταλαβαίνω γιατί τα συνδικάτα δεν έχουν πιο ενεργό ρόλο. Γιατί δεν τους ζητάτε να έχουν ένα πιο ενεργό ρόλο. Πιστεύω ότι αυτό θα έπρεπε να γίνει και θα ήθελα να προσθέσω και κάτι άλλο. Ε, στην εισαγωγή λέτε ότι αν έχουμε ε, υπερβολικές κανονισμούς και υπερβολική φορολόγηση, αυτό ενθαρρύνει την μαύρη εργασία. Με την πλατφόρμα αυτήν δεν αναφέρεται την, ε, την υπερβολική φορολογία και νομίζω ότι αυτό είναι μια αδυναμία. Θα πρέπει να συμπεριληφθεί σε αυτό και θα πρέπει να ρυθμιστεί η υπερβολική φορολογία. Ευχαριστώ λόγω στην κυρία Σοβιέσκα Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αναφίβολα η δηλώτη εργασία η ψευδής αυτοπασχόληση είναι τεράστιο πρόβλημα για την Ευρώπη και αν καταφέρουμε να το καταπολεμήσουμε θα αλλάξει πολύ κατάσταση. Είπατε ότι δεν υπάρχει συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη όμως θεωρώ ότι τέτοια συνεργασία υφίσταται ήδη. Υπάρχουν επιτροπές και ομάδες εργασίας που ε, ασχολούνται με την δήλωτη εργασία. Υπάρχουν επιθεωρητές οι οποίοι ασχολούνται με αυτό το θέμα. Υπάρχει επιτροπή ε, που ασχολείται με την απόσπαση των αποσπασμένους εργαζόμενους. Υπάρχει Επιτροπή Απασχόλησης, Διοικητική ε, Επιτροπή, Συντονισμού για την Κοινωνική Ασφάλιση. Υπάρχει επίσης μια ομάδα εργασίας για την διοικητική συνεργασία σε θέματα φορολόγησης και ε, σε αυτήν ε, περιλαμβάνεται και μια προσπάθεια ανταλλαγής πληροφοριών. Τα κράτη-μέλη ενδιαφέρονται να συνεργαστούν για την καταπολέμηση της ε, αδίλωτης εργασίας. Επομένως, η ερώτηση που θέλω να θέσω είναι δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους υπάρχοντες μηχανισμούς του, το σύστημα IMI. Έχουμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο ε, χρησιμοποιείται στην Ευρώπη και θεωρώ ότι η εμπλοκή των κρατών μελών στην ανταλλαγή πληροφοριών είναι πολύ επιτυχής. Ήδη μπορούμε να την επεκτείνουμε φυσικά. Έχουμε ηλεκτρονικό σύστημα ανταλλαγή πληροφοριών σε θέματα κοινωνική ασφάλιση και αυτό το εργαλείο μπορούμε να το αξιοποιήσουμε. Δεκατομμύρια χρειάζονται για να δημιουργηθεί αυτή η πλατφόρμα και αυτό με ενισχύει και συνέχεια 20.000 ευρώ προβλέπονται για έξοδο ταξιδίου κτλ. Πρέπει να καταπολεμήσουμε την αδειλωτή εργασία, αλλά με τον πιο αποδοτικό τρόπο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η αδήλωτη εργασία Υπάρχει ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι πρόβλημα, υπάρχει ε, φοροδιαφυγή, έλλειψη εισφορών κλπ. Αλλά έχουμε και αδικήματα, εγκληματικές πράξεις. Για όλα αυτά τα θέματα συμφωνούμε ότι πρέπει να υπάρξει νομοθεσία για να καταπολεμηθούν αυτά τα προβλήματα, ούτω ώστε αυτοί που καταχρώνται το φορολογικό σύστημα να προσάγονται στη δικαιοσύνη. Ωστόσο, θα πρέπει αυτή η νομοθεσία να θεσπιστεί από δημοκρατικά εκλεγμένους και πολιτικούς οι οποίοι λογοδοτούν σε εθνικό επίπεδο και όχι από το μη δημοκρατικό ευρωπαϊκό κοινοτικό επίπεδο. Έχουμε την πολιτική ανοιχτών θυρών ε, στο, στην Ευρώπη και αυτή η προτινόμενη νομοθεσία απλώς καταδεικνύει πόσο αυτή η πολιτική είναι ανέφικτη στην πράξη. Εάν 500 εκατομμύρια άτομα δεν είχαν το δικαίωμα να ζουν και να εργάζονται και να έχουν κοινωνικά, κοινωνικές παροχές στο Ηνωμένο Βασίλειο, τότε θα μπορούσαμε να αρχίσουμε να ασχολούμεθα με την ψευδή και ε, αδήλωτη εργασία, χωρίς ε, να αναμειγνύεται στους εσωτερικούς μας νόμους η Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι η νομοθεσία αυτή θα είναι η απαρχή ενός μιας αρπαγής εξουσίας, υφαρπαγής εξουσίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, που εμποδίζει τις εθνικές αρχές να έχουν ε, τους φορολογικούς τους νόμους. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι αποφασισμένο να σταματήσει οποιαδήποτε ενοποίηση, ελοκλήρωση αυτού του είδους. Ε, ενώ οι ψηφοφόροι δεν κατανοούν ότι αυτό έχει αρχίσει να συμβαίνει. Επίσης είμαι αντίθετη στο να ξοδευτούν 1,2 εκατομμύρια ε, για, ε, για ένα άλλο talking shop, ένα πλαίσιο συζήτησης για να συζητηθεί το θέμα αυτό. Επίσης, δεν έχετε αντιληφθεί ποια είναι η οικονομική κατάσταση σε πάρα πολλές οικονομικές χώρες χρειάζεται λιγότερη παρέμβαση, ε, λιγότερες ε, δαπάνες. Ε, εμείς θα ζητήσουμε να καταψηφιστεί αυτή η πρόταση και θα κάνουμε έκκληση σε όλους να πράξουν το ίδιο. Θα ήθελα να επανέλθει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ναι, με ιδιαίτερη χαρά Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να απαντήσω στα ερωτήματα των Ευρωβουλευτών, οι οποίοι είναι δημοκρατικά εκλεγμένοι, όσον αφορά τις παρατηρήσεις κυρίας Στάνρου, καταρχάς, και της κυρίας Ριμπέιρο, όσον αφορά τη θέση των κοινωνικών εταίρων στην πλατφόρμα αυτή. Πρέπει να πούμε δύο πράγματα. Πρώτον, από τη μία πλευρά έχουμε τους κοινωνικούς εταίρους σε επίπεδο ευρωπαϊκό, επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή, δηλαδή τις διάφορες ομοσπονδίες ή διακλαδικές ευρωπαϊκές οργανώσεις, οι οποίες όπως σας είπα έχουν ήδη καθεστώς παρατηρητή στην πλατφόρμα αυτή, όπως συμβαίνει άλλωστε και σε άλλα σχετικά φόρουμ, αλλά στα άλλα αυτά φόρα, σε αυτά που γνωρίζω τουλάχιστον, είναι ιδιαίτερα δραστήριοι οι παρατηρητές. Να επιστήσω επίσης την προσοχή των Ευρωβουλευτών στο άρθρο 5 της πρότασης, ένα άρθρο σημαντικό, άρθρο κλειδί, γιατί εκεί ζητάμε στα κράτη-μέλη να οργανωθούν κατά τέτοιο τρόπο, συνεκτικό δηλαδή και συντονισμένο, προκειμένου να είναι σε θέση να εργαστούν με τρόπο σφαιρικό και ολιστικό. Στο άρθρο αυτό επίσης προβλέπεται, ακριβώς επειδή γνωρίζουμε ότι σε εθνικό επίπεδο διαδραματίζεται ένα σημαντικός ρόλος από τους κοινωνικούς εταίρους και οι κοινωνικοί εταίροι βέβαια είναι οι εκπρόσωποι των εργοδοτών αλλά και των συνδικάτων. Υπάρχουν δηλαδή ορισμένα κράτη-μέλη τα οποία ήδη έχουν θεσπίσει πολύ αποτελεσματικές στρατηγικές είτε σε εθνικό είτε σε τοπικό επίπεδο, στρατηγικές συνεργασίες με τους κοινωνικούς εταίρους και βέβαια θα πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτές τις θετικές εμπειρίες. Μπορούν λοιπόν στα πλαίσια της πλατφόρμας αυτής ε, οι αντιπροσωπείες των κρατών μελών μπορούν να εντάξουν τους κοινωνικούς εταίρους οι οποίοι ήδη συμμετέχουν σε ανάλογες δομές σε εθνικό επίπεδο. Τώρα, όσον αφορά τα φορολογικά ζητήματα, πρέπει να σας πω ότι η πλατφόρμα αυτή μπορεί να εξετάσει την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα. Να σας υπενθυμίσω επίσης ότι ε, η πρόταση αυτή βασίζεται στο άρθρο 153 της συνθήκης, βάσει του οποίου οφείλουμε να εργαστούμε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που μας ε, δίνονται από αυτή τη νομική βάση. Να σας όμως επίσης ότι ε, η νομική αυτή βάση, η οποία προβλέπει την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέτρων υποστήριξης για να συμπληρωθεί η δράση των κρατών μελών. Η νομική λοιπόν αυτή βάση δεν προβλέπει ρυθμιστικά νομοθετικά μέτρα, αλλά ανταυτού προβλέπει τη δημιουργία μιας πλατφόρμας συνεργασίας με την εξαίρεση της εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας. Προφανώς η νομοθεσία παραμένει αρμοδιότητα εθνική. Τα κράτη-μέλη αυτά δηλαδή πρέπει από μόνα τους να νομοθετήσουν σε εθνικό επίπεδο λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της επιτόπου αγοράς εργασίας. Τώρα όσον αφορά το προπολογισμό της πλατφόρμας αυτής. Ο προπολογισμός είναι καθαρά ενδεικτικό στη φάση αυτή. Θα διαφέρει από τον ένα στο άλλο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντως εκτιμά ότι 2,5 εκατομμύρια ευρώ σε αιτήσια βάση για την διοργάνωση, σύνθεση της πλατφόρμας αυτής και για την υποστήριξη ορισμένων επιχειρησιακών μορφών συνεργασίας αρκούν. Επίσης με τα κονδύλια αυτά θα μπορούν πραγματικά οι εκπρόσωποι τα κράτη-μέλη να συνεδριάζουν για να συζητάνε για κάποιες κοινέ αρχές και είναι ένας προπολογισμός ο οποίος δεν θα έχει δημοσιονομική επίπτωση όσον αφορά τους προπολογισμούς των κρατών μελών. Ευχαριστώ. Θα ορίσουμε εισηγητή στις 4 Σεπτεμβρίου. Μερικές ακόμα παρατηρήσεις. Η ερώτηση που θέτε είναι αν αυτή η Επιτροπή θα συνεργαστεί με εμπειρογνώμονες και άλλες ενδιαφερόμενες φορείς πάνω σε αυτό το θέμα. Αν βοηθάει αυτή την πλατφόρμα στην καταπολέμηση της αδίλωτης εργασίας, τότε αυτό θα είναι καλό. Η αδίλωτη εργασία είναι ένα οργανωμένο έγκλημα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπό αυτή την έννοια είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε τις εργασίες μας επί του θέματος σε αυτή την Επιτροπή και να μπορέσουμε να είμαστε αποδοτικοί. Αυτά στο σημείο 5 της μερίσιας διάταξης. Ο λόγος στην Τανούτα. Θέλω να διευκρινίσω κάτι. Είπατε ότι το κόστος είναι 2,5 εκατομμύρια, το κόστος της πλατφόρμας αυτό είπατε. Θα ήθελα να καταλάβω ακριβώ τι είπατε. Είπατε ότι το συνολικό κόστος, είπατε ότι είναι 2,5 ευρώ ανά άτομο. Αυτό είπατε. Όχι είπα, ναι, ναι, ότι η Επιτροπή για να υποστηρίξει τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας είχε προβλέψει 2,5 εκατομμύρια κατέτος, είναι ένας ενδεικτικός μέσος όρος και είναι ένα λογικό ποσό σε σχέση με τα διακυβεύματα αυτού του θέματος της αδήλωτης εργασίας στην Ευρώπη. Okay, damit haben wir den Tagesordnungspunkt. Ολοκληρώσαμε και το σημείο 5. Πάμε στο 6. Επόμενες συνεδριάσεις. Πρωτόν να φερθώ στις ημερομηνίε. Να ευχαριστήσω τη Γραμματεία για την προετοιμασία της συνεδρίασης. Βλέπω τώρα ως πρόεδρος πόσο σημαντική είναι η εργασία τους. Ευχαριστεί και τους διερμηνείς ο Πρόεδρος. Έχετε καλό καλοκαίρι και καλή επιστροφή το Σεπτέμβριο με, γεμάτη με ενέργεια. Θα ξανασυναντηθούμε ε, και πάλι στις 3 Σεπτεμβρίου από τις 3 μέχρι τις 6.30 και στις 4 από τις 9 το πρωί ή 10 μέχρι τις 12. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Καλές διακοπές.